Μία μόνο αποχή. Ωραία. Ευχαριστώ. hier noch ein was abzustimmen haben von Evans. Äh, Βλέπω ότι μπορούμε να περάσουμε και στην επόμενη ψηφοφορία της ε, Jill Evans ηλεκτρονικά τέλος της ψηφοφορίας και εδώ εγκρίνεται βέβαια. 20. Περνάμε στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης. Ψηφίζουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε κυρία Κορόλα. Εγώ έχω ένα πρόβλημα με τη μηχανή μου, τεχνικό, δεν δουλεύει. Μπορείτε να ψηφίσετε δίπλα. Έχω ψηφίσει τρεις-τέσσερις φορές, αλλά δεν δουλεύει. Ο Κρίς. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς τι ψηφίζουμε. Ποια έκθεση ψηφίζουμε τώρα. Το 20, σημείο 20 στην ημερήσια διάταξη. Εχθές συζητήσαμε, όπως θυμάστε, στην Επιτροπή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτοί που ήταν εδώ το θυμούνται φαντάζομαι. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το σημείο 20. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 15 κατά, μία αποχή. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, το σημείο 21 της ημερησίας διάταξης. Για, την, ε, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, την φαρμακοεπαγρύπνηση. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 38 από κοινό ψηφίζουμε τις δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, όχι. Ωραία. Την 39 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στις 40, 41, 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 Α, όχι, ελέγχουμε την 40, 41, 42. Ψηφίσατε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 43 και 19 από κοινού όμως. Ε, συγγνώμη, και 90 από κοινού. Κατά αποχές. Με την ίδια ακριβώς πλειοψηφία. 44, 89. Α, όχι, επανερχόμαστε στην προηγούμενη ψηφοφορία και ελέγχουμε την 43 και την 90. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 44 και 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 και 91 μαζί. Όχι. Ναι. Ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48, 51, 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 μέχρι την 25 κατά αποχές απορρίπτονται. 52 κατά αποχές απορρίπτεται. Η 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 μέχρι 3 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 α όχι να ελέγξουμε την 9 έως την 3 ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι τέλος απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59-31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Κατά αποχές 62 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 μέχρι την 6. αποκτήτεται 50, ε, συγγνώμη, 65 υπέρ κατά απορρίπτεται. Α, να ελέγξουμε. 56 μέχρι την 105. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Ναι, έχουμε κάτι για την τέτοια. Κατά. Απορρίπτεται. 10 μέχρι 81 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 71. Το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται 72 σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται το δεύτερο υπέρ κατά το δεύτερο α καταπίπτει 73 υπέρ κατά απορρίπτεται 74 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Α, να ελέγξουμε την 74. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 74. 75. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Την ελέγχουμε κι αυτήν. 75 ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται 75. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά βοχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 79 και 80. Α, όχι. Ελέγχουμε την 78. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 79 και 80 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαναλαμβάνουμε ηλεκτρονικά 79 και 80. 79 και 80. Τέλος. Εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Όχι, καταπίπτει 82. 83 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 84. 85 κατά 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 με μία προφορική υποτροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε με την προφορική υποτροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στα παραρτήματα. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85. Α, συγγνώμη. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Ναι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Α, καταπίπτει. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 109. 110 μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικά. Την 109-110. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Ωραία. Και τώρα πάμε στην 15, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 16, υπέρ, Α, θέλετε να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την προηγούμενη. Ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 και 24 μαζί υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά την 23 και 24 ψηφίσατε Τέλος. Απορρίπτεται. 25. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της 25. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποχές. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο του κειμένου. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Μία αποχή μόνο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Μία αποχή. Συγχαρητήρια. Λίντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Και επειδή πρόκειται για κάτι τεχνικό, πρέπει πραγματικά να αρχίσουμε να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί στο θέμα της φαρμακοεπαυρίκησης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό που κάναμε σήμερα. Και βεβαίως ε, εδώ χρειαζόμαστε να δοθεί εντολή. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Λείπουν τρεις ψήφοι. Δύο λείπουν. Τέλος. 44 υπέρ, ένας κατά. Είμαστε εντάξει με την εντολή και σας εύχομαι και καλή επιτυχία. Έτσι κι αλλιώ ε, η Λίντα Μαγκιάβινγκ δεν έχει τίποτα να κάνει. Ολοκληρώθηκε η αποστολή της. Οπότε ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Αυτοί που θέλουν να φύγουν, να φύγουν καλά Χριστούγεννα και ελπίζω το 2014 να είναι καλό. Σας εύχομαι υγεία, χαρά και εις το επανειδήν. Πραγματικά σας εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά εμείς θα συνεχίσουμε εδώ με την επόμενη έκθεση, την έκθεση του Πίτερ Λίζε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι βεβαίως πρέπει να συνεχίσουμε. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας είχε απασχολήσει εδώ και χρόνια με διαφορετικές πτυχές και θα ήθελα καταρχήν να σας υπενθυμίσω πού βρισκόμασταν και γιατί μας απασχολεί σήμερα το θέμα αυτό. Να σταματήσετε όμως τις διμερείς σας συζητήσεις, διακόπτω για λίγο. Για σφυρελατίστε λίγο κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να ηρεμήσετε λίγο, χρειάζεται ησυχία για να μπορέσουμε να προσέξουμε και να ακούσουμε τον Πίτερ Λίζα. Κυρία Γιανακουδάκη. Κυρία Γιανακουδάκη, μήπως μπορείτε Πίτερ, έχεις το λόγο. Λοιπόν, όλοι αυτοί που έχετε να κάνετε κάποια άλλα πράγματα, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, γυσμένο το καινούριο χρόνο και εμείς θα ασχοληθούμε εδώ με τις αερομεταφορές και τις εκπομπές οι οποίες αυξάνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της, ε, του ΙΚΑΟ, του Διεθνούς Οργανισμού για την πολιτική αεροπορία, βασιζόμαστε στα στοιχεία που έχουμε, που φτάνουμε τα 900 τόνους. 900, 900 εκατομμύρια τόνους, συγγνώμη. Μπορούμε εδώ να συγκρίνουμε με τα προηγούμενα στοιχεία που έχουμε και τα σενάρια είναι φυσικά ότι αυξάνονται και το 2015 θα έχουμε ακόμα μια αύξηση της τάξης του 20% και βεβαίως οι προσπάθειες που γίνονται σε άλλους τομείς για τον περιορισμό των εκπομπών και τις αρνητικές επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίματος θα πρέπει βεβαίως και να μας απασχολήσουν στον τομέα των εκπομπών που προέρχονται από τις αεροπορικές μεταφορές. Ήδη από το 1992 έχει αρχίσει ο ΙΚΑΟ να ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό και φυσικά το θέμα των εκπομπών που προέρχονται από τον τομέα των αερομεταφορών και τον περιορισμό αυτών των εκπομπών δυστυχώς δεν είχε μέχρι τώρα σημαντικό αποτέλεσμα. Εδώ και δέκα χρόνια πρέπει να σας πω μετά την συνάντηση στο Κιώτο δεν υπάρχει διεθνή συμφωνία υπογεγραμμένη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιες πρωτοβουλίες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 90% στήριξη είχαμε υποστηρίξει και στο Συμβούλιο πρέπει να σας πω ότι πέρασε ομόφωνα αυτή η πρόταση. Με το θέμα βεβαίως της συμμετοχής τρίτων κρατών σε αυτές τις συμφωνίες, η νομική τους οποίους ε, διαβουλευτήκαμε έχουν γνωμοδοτήσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο σαφώς και χρειάζεται την στήριξη των τρίτων χωρών, κάτι που είναι συμβατό με τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Υπάρχει σήμερα όμως παρόλα αυτά σημαντικό πρόβλημα με την αύξηση των εκπομπών και βεβαίως από την άλλη βλέπουμε σε τρίτες χώρες, να υπάρχει σημαντική στήριξη επιδοτήσεις των αερομεταφορέων και παραδείγματος χάρη για την εταιρεία Ryanair βλέπουμε ότι το 2012 η επιβάρυνση για αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία ήταν 0,03. Δηλαδή μιλάμε για ένα πάρα πολύ ε, χαμηλό ποσό, άλλες εταιρείες επιβαρύνονται λίγο παραπάνω. Απλώς σας το λέω για να καταλάβετε γιατί ποσά μιλάμε. Πρόκειται για cents. Σπάνια τα ποσά αυτά φτάνουν ε, τα ευρώ. Στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχει ένα τέλος, ένα τέλος που επιβαρύνει περισσότερο τις αεροπορικές εταιρείες, τις Ηνωμένε Πολιτείες Έχουμε 16,3 δολάρια επιβάρυνση για τις αεροπορικές εταιρείες που μεταφέρουν επιβάτες. Περίπου 2,5 δολάρια είναι ο μέσος όρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για πολύ χαμηλά ποσά και όταν ε, βεβαίως θεσπίστηκε αυτό το σύστημα για την ε, εμπορία των εκπομπών τα ποσά που αποφασίστηκαν, που βεβαίως ε, εξαρτώνται από τη διαδρομή, από τη χώρα υπέρπτυσης και σας επαναλαμβάνω ότι ο τρόπος υπολογισμού αυτών των τελών, αυτών των επιβαρύνσεων, οδηγούν σήμερα σε κάποια ποσά και εδώ βασίστηκα στο γερμανικό και στο βρετανικό σύστημα που βλέπουμε ότι βεβαίως έχουν κάποια επίπτωση αλλά αν συγκρίνει κανείς τι γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως σε τρίτες χώρες δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό το σύστημα. Τι κάναμε λοιπόν πέρσι. Η οδηγία τροποποιήθηκε μόνο για το 12 συγκεκριμένα και ξαναείδαμε όλες τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα που θέλαμε να πετύχουμε, ο στόχος κατά την άποψή μου δεν είναι πάρα πολύ φιλόδοξη. Εν αυτή ήταν η συμφωνία που επετεύχθη και ελπίζω Ελπίζουμε όλοι ότι αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα, μικρό βήμα πρόοδου. Πρέπει να σας πω ότι οι συνομιλίες που είχαμε με τις αρχές του ΙΚΑΟ οδήγησαν σε κάποιες βελτιώσεις και κατά κάποιο τρόπο εκπλήσωμε γιατί οι ίδιοι οι οποίοι επικρίνουν την έλλειψη αποτελεσμάτων στη Σύνοδο της Βαρσοβίας παραδείγματος χάρη, οι ίδιοι, οι ίδιοι που πραγματικά ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή, οι ίδιοι όταν μιλάμε για επιβάρυνση των αεροπορικών εταιριών, θεωρούν ότι αυτά που έχουν γίνει και αυτά που έχουν αποφασιστεί αρκούν. Οι στόχοι που έχουν τεθεί μέχρι τώρα είναι μέχρι το 2020 και σκοπός βεβαίως είναι μια πολύ δραστική, πολύ σημαντική μείωση των εκπομπών μετά το 2020, για την περίοδο μετά το 2020. Και στον ΙΚΑΟ δεν υπάρχει καμία μέχρι τώρα πρόταση και συζήτηση για περιορισμό των εκπομπών έως το 2020. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Μέχρι σήμερα η πρόταση είναι όχι αύξηση, αλλά δεν μιλάμε ακόμα για μείωση για την περίοδο μέχρι το 2020. Εγώ θα ήθελα να χαρακτηρίσω όλη αυτή την πρόταση σαν απογοητευτική. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε καταρχήν να πιέσουμε περισσότερο και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις λίγο πιο αποτελεσματικές για το 2000, μέχρι το 2020. Σήμερα υπάρχουν πολλοί, όπως παραδείγματος χάρη οι εκπρόσωποι των εταιριών low cost, η... ο φορέας που τους εκπροσωπεί είναι η ΕΛΦΑ, θεωρούν ότι τα πράγματα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν και ότι δεν πρέπει να υπάρξει απολύτως καμία αλλαγή. Άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει αυτή η οδηγία stop the clock να επεκταθεί για ένα έτος. Η πρόταση τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια συμβιβαστική πρόταση, ξεκάθαρα. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, θα πρέπει οι διαδρομές αυτές να συνεχίσουν να συνυπολογίζονται μέχρι το 2020 και αυτό όχι μόνο εάν απογειώνονται και προσγειώνονται στην Ευρώπη, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ακόμα και αν απλώς υπάρχει μια υπέρπτυση. Παραδείγματο χάρη μια πτήση από το Λονδίνο στην Αθήνα, αλλά και τις πτήσεις που όπως ξέρετε υπάρχουν όλο και περισσότερες πτήσεις που περνάνε από το αεροδρόμιο της Κασταντινούπολης. Η οποία έχει, το αεροδρόμιο αυτό έχει αποκτήσει τεράστια, τεράστιο αριθμό πτήσεων. Για μένα λοιπόν αυτό είναι μια φιλόδοξη αλλά απαραίτητη πρόταση. Θα πρέπει πραγματικά να δούμε και οι σύντομοι υπολογισμοί που κάναμε μέχρι τώρα μας δείχνουν ότι θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερος περιορισμός των εκπομπών εάν περάσει αυτή η πρόταση. Προς το παρόν ε, συζητούμε μόνο αντισταθμίσματα και βεβαίως ε, εδώ το σύστημα έτσι όπως έχει καταρχήν ε, αρχίσει η επεξεργασία είναι για σταθεροποίηση για τα ποσά τα οποία θα πρέπει να καταβάλουν ε, οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά βεβαίως ε, αναφερόμαστε και πολύ συγκεκριμένα και για μια μείωση από εδώ και πέρα των εκπομπών. Όπως ξέρετε, πολλοί επικαλούνται στρέβλωση του ανταγωνισμού και μάλιστα υπάρχει και το θέμα της προσφυγής στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Αλλά πραγματικά το παράδειγμα του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης που επαναλαμβάνω έχει αποκτήσει τεράστια σημασία το οποίο η κυκλοφορία αυξάνεται διαρκώς. Εκεί υπάρχει πραγματική στρέβλωση του ανταγωνισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί κάθε φορά που συνάντησα εκπροσώπους ε, τρίτων χωρών δεν ε, επικαλούνται νομικό ε, πρόβλημα. Κανείς δεν επικαλείται σήμερα ότι η πρόταση της Επιτροπής εμπεριέχει νομικές δυσκολίες. Το Συμβούλιο του ΙΚΑΟ και όλοι οι εκπρόσωποι της πολιτικής αεροπορίας το Συμβούλιο το δέχτηκαν. Σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση, αλλά αυτό είναι πολιτικό θέμα, δεν είναι νομικό. Και βεβαίως όπως ξέρετε μια τέτοια απόφαση όπως το stop the clock μπορεί να μην είναι δεσμευτική. Η απόφαση, όπως ξέρετε, του ΙΚΑΟ επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με την απόφαση του ΙΚΑΟ μία πτήση από τη Φραγκφούρτη στο Λονδίνο εμπίπτει αλλά το θέμα των τρίτων κρατών ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Λοιπόν, τι προτείνω εγώ τώρα σαν τροπολογίες. Μια πολύ βασική και ουσιαστική τροπολογία και νομίζω ότι εδώ είναι συμβαστικές οι προτάσει που κάνουμε γιατί υπήρχαν αρκετά ακραίε ε, ε, τοποθετήσεις είναι η πιθανή επαναεπεξεργασία του κειμένου πριν το 2020 και βεβαίως ε, ένας κανονισμός ε, που θα πρέπει να ισχύει μετά το 2020. Προσαρμογή λοιπόν της νομοθεσίας μας εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί εδώ για θέματα προτεραιότητας, όχι μόνο για τη δική μας Επιτροπή, αλλά και για την Επιτροπή των ε, Μεταφορών, είναι το θέμα των μέσων, καθώς και τη δυνατότητα προαιρετικής ε, εφαρμογής. Οι Υπουργοί Οικονομικών ε, των κρατών μελών έχουν εδώ κάποιες προτάσεις, αλλά πραγματικά η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών, σύγχρονων τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον που δεν επιβαρύνουν το κλίμα είναι κάτι που σαφώς θα πρέπει να υποστηριχθεί. Θεωρώ ότι οι επικρίσεις των τρίτων χωρών δεν πρόκειται βεβαίως να σταματήσουν από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχουν και όλες οι οικονομικές επιπτώσεις αλλά πραγματικά ο εναέριος χώρος ε, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα σημεία που θα πρέπει να, ε, στα οποία δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε. Η θέση του Κοινοβουλίου επίσης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη όσον αφορά την ίση μεταχείριση αυτών των τομέων, γιατί προς το παρόν βλέπουμε με σαφήνεια ότι είμαστε πολύ πιο ελαστικοί θα έλεγα στην εναέρια κυκλοφορία σε σχέση με άλλους τομείς στις διαπραγματεύσεις σας με τις ε, τρίτες χώρες και στις ε, προαιρετικές ε, εφαρμογές κάποιων διατάξεων ή στις εξαιρέσεις. Με τους συντονιστές συζητήσαμε και τα σημεία τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν στον τριμερή διάλογο, πριν ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος. Και βεβαίως όσον αφορά αυτό το stop the clock, οι πληροφορίες που έχουμε βάσει των στοιχείων του 2012 και επαναλαμβάνω εδώ περιοριζόμαστε μόνο στην ενέργεια κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας δείχνουν ότι σήμερα υπάρχουν ε, κράτη που δεν έχουν ακόμα απαιτήσει όλα τα πιστοποιητικά από εταιρείε εταιρείες για το 2012. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μας ε, αποδυναμώνει αποδυναμώνει τα στοιχεία, πολλές φορές δεν είναι πλήρη. Εμείς, σε περιπτώσει, για το 2012 είχαμε συμφωνήσει σε, μια, σε ένα κατώτατο όριο, σε μια ελάχιστα αποδεκτή λύση. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια. Και μέχρι τις 30 Απριλίου θα πρέπει εδώ να ληφθεί απόφαση βάσει στοιχείων που ελπίζω να είναι πλήρη. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να αποφασίσουμε, αλλιώς, αλλιώς επαναλαμβάνω στις 30 Απριλίου θα ληφθεί απόφαση ερήμην μας, χωρίς να μπορούμε να επηρεάσουμε. Ελπίζω λοιπόν να βρεθεί η συμβαστική λύση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε την μάχη. Θέλουμε τα, οι τρίτες χώρες να ε, συμμετάσχουν, θα ακούσουμε τα επιχειρηματά τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα εγκαταλείψουμε την μάχη. Εγώ πραγματικά ακούω τους εκπροσώπους των αεροπορικών εταιριών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν εμείς ασκούμε πίεση στους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αεροπορικών μεταφορικών εταιριών και ε, κατόπιν βλέπουμε ότι οι εταιρείες των τρίτων χωρών δεν υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις, όντως εδώ υπάρχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και αυτό βεβαίως και από μέρους των κρατών μελών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πραγματικά να έχουμε μία ενιαία τοποθέτηση, να είμαστε ενωμένοι έτσι ώστε να μπορέσουμε να βαρύνουμε όταν ε, διαπραγματευόμαστε με την Κίνα και τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές, περνάμε από λίγα ευρώ σε 40 παραδείγματος χάρη είναι αυτό που επιβάλλει η Γερμανία. Θα πρέπει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε μια κοινή πρόταση γιατί αυτό θα ενισχύσει την θέση μας. Συνομιλούσα με, μια, με τον εκπρόσωπο μια, μια σημαντικής αεροπορικής εταιρείας για τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα και βεβαίως εκεί προέκυψε και το θέμα άλλων πολιτικών ε, αν θέλετε πτυχών των συζητήσεων, όπως παραδείγματος χάρη τα ανθρώπινα δικαιώματα, το θέμα του Δαλάη Λάμα. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν πρέπει να ε, αποδυναμώσουμε τη θέση μας και να υποχωρήσουμε γιατί η Κίνα μας απειλεί. Οι αρχές μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εδώ να αποδυναμωθούν και καταλαβαίνετε ότι και οικονομικά και πολιτικά θα πρέπει να είμαστε ισχυροί. να μπορούμε να συνεχίσουμε από κοινού σε όλα τα μέτωπα να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, να δούμε πού μπορούμε με την Κίνα ή με τις Ηνωμένε Πολιτείες να αναπτύξουμε κοινά προγράμματα, κοινά σχέδια, αλλά σε καμία περίπτωση το θέμα της πίεσης από τις τρίτες χώρες να είναι το μοναδικό επιχείρημα ενός Ευρωπαίου νομοθέτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ πολύ τον Πίτερ Λίζε. Για τους σοσιαλιστές, ο σκιώδης εισηγητής είμαι εγώ και θα ήθελα να στηρίξω αυτό που είπε ο Πίτερ Λίζε. Είναι θέμα αρχής αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβληθεί ένα τέλος, ένας φόρος όπου θα είναι πολύ πιο ε, υψηλό από αυτά που προβλέπει το σύστημα ανταλλαγής ε, των εκπομπών. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σήμερα υπάρχουν μικρές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες κάνουν παραδείγματος χάρη διαδρομές και πτήσεις μεταξύ των νησιών και την ίδια ώρα έχουμε τον ε, μεγάλο αερομεταφορέα που κάνει μια πτήση μεταξύ Λονδίνου και Ουάσιγκτον και τα φορολογικά κίνητρα, αν θέλετε η φορολογική ε, κατάσταση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό την κατάσταση και πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί και να είμαστε σαφείς γιατί από τη στιγμή που όλοι αποφασίσαμε ήδη από το 2008 ότι οι αερομεταφορές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύστημα εμπορίας και ε, συναλλαγών των εκπομπών δεν πρέπει να ε, υποχωρούμε επειδή υπάρχουν αυτές οι πιέσεις. Επίσης με μεγάλη πλειοψηφία είχαμε πει ότι αυτό το stop the clock θα πρέπει να προχωρήσει και στις 30 Απριλίου το σύστημα που αποφασίσαμε θα πρέπει να, που, το, το παλιό μας σύστημα θα πρέπει να επανέλθει και να <coughs> λειτουργήσει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ έρχεται με μία νέα πρόταση, η οποία έχει νόημα. Είναι συμβιβαστική, είναι λογική και προσπαθεί να αποφύγει στρεβλώσεις ανταγωνισμού. Έχει δίκιο ο Πίτερ όταν αναφέρεται σε αυτό. Το θέμα είναι τι γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Θεωρώ λοιπόν λογικές αυτές τις προτάσεις και γι' αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή. Έχει νόημα και από άποψη αν θέλετε, περιβαλλοντολογική, αλλά όχι μόνο. Αν κοιτάξει κανείς τα οικονομικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν σήμερα τον κλάδο των αερομεταφορών, έχει νόημα αυτή η πρόταση. Τώρα, το θέμα του Δαλάη Λάμα. Πρέπει να ζητήσουμε συγνώμη από τους Κινέζους, επειδή τον συναντήσαμε. Πραγματικά, σαν Ευρωπαίοι, Είμαστε κυρίαρχα κράτη και νομίζω ότι είμαστε σε θέση να επιλέξουμε και να υποστηρίξουμε και τις επιλογές μας. Λοιπόν, σαφώς και όπως προτείνει ο Πετελίζη, σε κάποιες περιπτώσεις εδώ ζητάμε αυξήσεις της τάξης του 40-50% στα ποσά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε, να θεωρήσουμε ότι ο τομέας ε, της ενέργειας κυκλοφορίας είναι εξαίρεση. Οι επιπτώσεις ε, στις αλλαγές του κλίματος δεν μπορούν να ε, θεωρήσουμε ότι δεν επηρεάζονται από τις αερομεταφορές. Και βεβαίως σε διεθνές επίπεδο μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ τις επιδόσεις μας με πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα πρέπει να επιβληθούν όταν διαπραγματευόμαστε σε διεθνές επίπεδο. Τώρα, ο χρόνος πιέζει. Επαναλαμβάνω ότι στις 30 Απριλίου θα σταματήσει το σύστημα Stop the Clock και αν δεν κάνουμε τίποτα θα επανέλθει το προηγούμενο σύστημα, η παλιά νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν σίγουρα να δείξουμε πνεύμα συμβιβασμού. Αλλά επαναλαμβάνω μην ξεχνάτε ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, αν δεν βρούμε λύση, μετά τις 30 Απριλίου επανέρχεται το παλιό σύστημα. Και το θέμα είναι τι αποφάσισε ο ΙΚΑΟ για την πολιτική μετά το 2020. Ας προετοιμαστούμε λοιπόν για την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου Επαναλαμβάνω ότι εγώ υποστηρίζω την πρόταση του Πίτερ Λίζε και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι τρίτες χώρες να μας απειλούν και εμείς να υποχωρούμε. Είμαστε ανοιχτοί για διαπραγματεύσεις, αλλά είμαστε 28 κυρίαρχα κράτη και θα πρέπει να μην διασπαστούμε αλλά να σταθούμε ενιαίοι και δυνατοί στις τοποθετήσεις μας. Επαναλαμβάνω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι υποστηρίζω την πρόταση του Πίτερ Λίζε. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν με τους άλλους σκιώδεις εισηγητές. Ο Chris Davis για τους φιλελεύθερους έχει το λόγο. Thank you very much, uh, Chairman. Um... ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω και θεωρώ ότι θα πρέπει οι αεροπορικέ εταιρείε να συμβάλλουν και αυτή στην αντιμετώπιση των ε, εκπομπών θερμοκηπίου Πολύ καιρό παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος. Φυσικά και αν επιτευχθεί συμφωνία αυτό θα είναι το πιο θετικό. Δεν ξέρω αν θα αποσπάσουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Δεν είναι στον εταιρεών και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να αναγκάσει, να πιέσει και άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, ούτως ώστε να αναλάβουν δράση. Βέβαια, για τις ευρωπαϊκές εταιρείες δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αν εμείς ε, μόνο μερός κάνουμε κάτι ως Ένωση, όπως τα είπε ο Πίτερ, και επομένως θα πρέπει να προωθηθεί αυτή η πρόταση του να χρεώνουμε μόνο τα δρομολόγια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θεωρητικά είναι θεμητό επιχείρημα, αλλά τι γίνεται όταν δεν πληρώνουν αυτό που πρέπει να πληρώσουν. Γιατί ξέρουμε ότι σήμερα δεν πληρώνουν. Και η διαδικασία παρακολύεται. Θα πρέπει επομένω τα κρατημήλια να φροντίσουν να εισπράττουν αυτά που πρέπει. Δεν κάνουν το κάνουν ε, σήμερα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να φύρουμε να μας ε, απειλεί η Κίνα, το Airbus κλπ. Και, και να αποφασίσουμε μέχρι πού θέλουμε να φτάσουμε όσον αφορά τις συνέπειες που θα υπάρξουν τι εμπορικές κλπ. Εάν επιμείνουμε στο να θέλουμε να υπάρχουν επιπληρωμές κλπ. Εγώ είμαι υπέρ του να χρεώνουμε τα δρομολόγια στον ενιαίο χώρο μας. Όμως να μην κάνουμε μετά πίσω, γιατί αυτό θα είναι ταπεινωτικό. Έτσι δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό με προβληματίζει. Επί της αρχής συμφωνώ. Οπότε να ακουστεί νέα η φωνή μας, ότι θα τα καταφέρουμε, είμαι υπέρ, 100%, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα τα καταφέρουμε. Και άλλο το ερώτημα είναι, εάν θα ρισκάρουμε ή όχι και να πούμε ότι θα προχωρήσουμε προς τα εκεί ή να θεωρήσουμε ότι μπορεί να μην τα καταφέρουμε εκ των προτέρων Οπότε με αυτή την πιθανότητα στο μυαλό ας είμαστε πιο, α, πιο, πιο προσεκτικοί. Αν βλέπω τον συνάδελφο. Γιατί δεν, ξέρω, τι θα κάνουμε. Ε, μέχρι σήμερα δεν τα έχουμε πάει και τόσο καλά σε αυτό το θέμα. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Πίτερ Λίζε για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Εξαιρετικά καλογραμμένη η έκθεση του και ιδιαίτερα η αιτιολογική έκθεση. Λυπάμαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό έχει υποχωρήσει εξαιτίας πολιτικών πιέσεων. Όπως είπαν οι συνάδελφοι, το αρχικό σύστημα ε, εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής έχει χαρακτηριστεί νόμιμο και αυτό δεν αλλάζει από οποιαδήποτε από οποιοδήποτε ψήφισμα του ΙΚΑΟ ή μέσω οποιασδήποτε πίεση από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όπως είπε ο κ. Λίζα άλλωστε, τα παράπονα περί υψηλού κόστους ε, είναι άχρηστα και αβάσιμα. Ε, τα άλλα τέλη είναι πολύ περισσότερα από ότι ε, τα τέλη εκπομπών που προβλέπει το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης συμφωνώ με τον Πίτερ Λίζε, οι κυβερνήσεις δεν είναι συνεπείς. Παραπονιούνται για πολύ μικρή πρόοδο στις χερσές μεταφορές, από την άλλη μεριά στις ενεργές μεταφορές αφήνουν τις αεροπορικές εταιρείες να κάνουν ό,τι θέλουν. Πόσο είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η συνέπεια, αναρωτιέμαι. Εν πάση περιπτώσει, η αύξηση των εκπομπών στην, ε, στις μεταφορέ μεταφορές είναι πολύ ψηλή, πολύ μεγάλη και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός αυτό. Η Κομισιόν αποφάσισε να επαναχωρήσει σε ένα μεγάλο βαθμό εξαιτία πολιτικών κριτικών που δέχτηκε, πολιτικών επικρίσεων που δέχτηκε. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι στην πρόταση του Πίτερ Λίζε έχουμε πολλά θετικά στοιχεία. Τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων θα πρέπει να διατίθενται ε, στην καταπολέμηση της ε, αύξησης θερμοκρασίας του πλανήτη και δεύτερον ε, θα πρέπει να δεχτούμε μια αναβολή έτσι ώστε ο ΙΚΑΟ να πάρει μια απόφαση αλλά όχι πολύ μεγάλη. Μετά από κάποια χρόνια, λίγα, θα πρέπει να επιστρέψουμε στο αρχικό μας σύστημα. Αυτό είναι το ελάχιστο. Τώρα, Οι πράσινοι πιθανότατα θα προτείνουν και ενίσχυση των προτάσεων του Πίτερ Λίζε, για παράδειγμα. Και ό,τι αφορά τις θάλασσες. Η περιοχή που καλύπτεται από το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών τουλάχιστον αποκλειστικές οικονομικές ζώνες σε ό,τι αφορά τις θάλασσες. Τα 12 ναυτικά μίλια είναι πολύ μικρή περιοχή, μικρή ζώνη, περιορισμένη. Επίσης, θα πρέπει να δούμε το μέγιστο όριο των εκπομπών και να αυξήσουμε το ποσοστό των πληστηριασμών όταν αφόσον μειώνεται η κάλυψη σε σχέση με την αρχική πρόταση. Όπως σας είπα ήδη, ορισμένες χώρες είναι ασυνεπείς. Μία εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι ένας φόρος επί των καυσίμων για τα αεροπλάνα, κάτι που θα είχε ισοδύναμα αποτέλεσματα. Όμως η νομοθετική διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί για τέτοιου είδους φόρο είναι πολύ πιο σύνθετη. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει υποστήριζοντας την αρχική πρόταση, την αρχική νομοθεσία Και επίσης το ότι οποιαδήποτε μείωση της κάλυψη θα πρέπει να είναι προσωρινή. Μάρτιν Κέλεμαν. Ευχαριστώ πολύ. Κέλεμαν. I don't normally like saying this because it destroys my credibility, but I think I generally agree with Chris Davis. Γενικά, δεν νομίζω ότι με περιποιεί τιμή, την αξιοπιστία μου την αναβαθμίζει, αλλά σε αυτή την περίπτωση συμφωνώ με τον Chris Davis, γιατί αυτό που είπε ο Μαρτίας και ο Πίτερ πρέπει να απαντήσουν σε ένα ερώτημα. Ακριβώς όπως εξήγησαν είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να ε, υπερασπιστούμε τις αρχές μας, είναι θέμα ευρωπαϊκών προτύπων, τέλος πάντων τελικά είναι πενταροδεκάρες και δεν κάνει μεγάλη διαφορά, είναι ένα-δύο ευρώ αναπτύσσει, άρα ας αναρωτηθούμε γιατί θέλουμε τότε να κάνουμε μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια γιατί να τα χαλάσουμε με τους ε, εταίρους μας Ινδία, Αμερική, δεν με νοιάζει για την Κίνα για κάτι που δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα. Επίσης θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα της μη συμμόρφωσης είτε σας αρέσει είτε όχι τελικά το πράγμα καταλήγει κάποιες χώρες ε, η Γερμανία, η Αγγλία με τη Φραγκφούρτη και το Χήθρο να έχουν κάποιες εταιρείε που δεν πληρώνουν. Και πολλές φορές αυτό ε, γίνεται και με την άδεια του νόμου. Δηλαδή ε, βλέπετε πόσο τις είναι οι κυβερνήσεις να εισπράξουν. Επομένως αυτά που λέμε δεν μπορείτε να γίνουν όπως είπε και ο Κρίς. Γιατί να θεωρούμε ε, ότι είναι τέτοιο θέμα Αρχίζει να μην ξέρουμε θα το πετύχουμε και τελικά αν μπορούν τα κράτη-μέλη, θα βρουν έναν τρόπο να μην συμμορφωθούν. Και νομοθετικά δεν θα το εφαρμόσουν. Άρα θα καταλήξουμε να ταπεινωθούμε. Εκεί θα καταλήξουμε με αυτή την πορεία που ακολουθούμε. Επομένως, ε, όπως και το 2013 να το 2020 και να δούμε τι θα γίνει το 2016 από τη συνέλευση της ΙΚΑΟ ε, και οπότε αναλόγως βλέποντας και κάνοντας με το 2016. Επομένως, αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια πρόοδο, να έχουμε κάποιο καθεστώς που να ισχύει παγκοσμίω και να μην δημιουργούμε ε, εντάσεις και συγκρούσεις από κάπου δεν είναι τόσο σημαντικό από πλευράς οικονομικής. Γιατί ξέρετε πόσο εχθρική, πόσο αρνητική είναι η στάση των χώρων μελών για αυτό που θέλουμε να χρειώσουμε. Άρα να γίνει μια συνολική συμφωνία για τι μεταφορές και αυτό θα πρέπει τελικά να επιδιώξουν. Πρόσοχη να μην διαταράξουμε τις χώρε με αυτούς τους εταίρου μα και ιδίω με τις ΗΠΑ. Γιατί αυτό θα γίνει. Και έχει σοβαρή ανησυχία για το τι θα γίνει με αυτή τη μη συμμόρφωση. Και με άλλε χώρες υπάρχει πρόβλημα. Και πολλοί επαγγελματικοί βιομηχανικοί κύκλοι θεωρούν ότι αυτό θα γίνει. Με αυτά τα οποία θέλουμε να συμφωνήσουμε ως, ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη κατά μόνας στα πλαίσια της ΕΚΑΟ. Είναι το θέμα βέβαια του περιβάλλοντος, το θέμα της τρέβλωσης του ανταγωνισμού, όλα αυτά θα είναι έτσι βλαβή για τις αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης και γενικά για το ΣΕΔΕ όλα αυτά θα είναι αρνητικά όλο το σύστημα θα το διαταράξουμε, θα το υπονομεύσουμε. Αν δεν συμφωνήσουμε μέχρι τον Απρίλιο, τότε το ΣΕΔΕ θα ξαναγυρίσει εκεί που βρισκόταν πριν από ένα-δύο χρόνια και ξέρετε ποιες είναι οι συνέπειες. Θα έχουμε αντίπεινα, πολιτικά, οικονομικά, από τρίτες χώρες. Άρα, Ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και κάτι τελικά να συμφωνήσουμε για, τις, ε, για αυτές τις τροπολογίες και βεβαίως να έχουμε και ένα εναλλακτικό σχέδιο εάν δεν τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη ακούσαμε, είπαν άλλοι. Να σας υπενθυμίσω ότι πριν από έξι χρόνια είχαμε προσπαθήσει να συμπεριλάβουμε σε αυτή τη συζήτηση και τις αεροπορικές εταιρείες. Από την πρώτη μέρα αυτής της προσπάθειας είδαμε πόσο δύσκολο ήταν να συμμετέχουν ε, οι τρίτες χώρες και βεβαίως οι διαμαρτυρίες έχουν ακουστεί, έγιναν ε, συζητήσεις ε, με το Συμβούλιο και τα παράπονα αυτών που δεν συμμετείχαν ακούστηκαν με πάρα πολύ ε, δρυμή τρόπο. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αυτή την πρόταση, αλλά αν ε, δει κανεί τα έγγραφα του ΙΚΑΟ, πριν το Σεπτέμβριο διαβάζω, γιατί κοίταξα πολύ προσεκτικά αυτά τα και υπήρχαν άντρα που αναφερόταν στη στάση των τρίτων χωρών, στα μέτρα που ενδεχομένως ε, θα μπορούσαν να δεχτούν ή όχι και πρέπει να σας πω ότι στον ΙΚΑΟ έγινε ψηφοφορία με πολύ, πολύ οριακό αποτέλεσμα. Αυτό είναι σπάνιο στον ΙΚΑΟ και γι' αυτό και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία προκάλεσε αυτές τις ε, προτάσεις. Επαναλαμβάνω, η στάση των τρίτων χωρών δεν νομίζω θα αλλάξει. Το θέμα δεν είναι από νομικής απόψεως ε, ποιος έχει δίκιο. Φυσικά και εμείς έχουμε δίκιο. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, το νομικό σύστημα, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να επιβληθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ δεν είναι έξυπνο να επιμένουμε σε αυτό το μοντέλο. Διότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί απλούστατα. Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε εκτός. Και δεν είναι θέμα κόστους. Ε, έχει δίκιο ο Ματίας όταν αναφέρεται σε θέματα αρχών. Το θέμα είναι ποια είναι η αρμόδια αρχή, ποιος αποφασίζει, ποιος μπορεί να επιβάλλει ένα τέλος. Το θέμα αυτού του μοντέλου αέριου χώρου εμείς μπορούμε να το στηρίζουμε. Αλλά πραγματικά το λιγότερο που θα έπρεπε κανείς να σκεφτεί πριν να το υποστηρίξει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ποιοι άλλοι το δέχονται. Θεωρώ λοιπόν ότι ίσως θα ήταν πιο έξυπνο να συνεχιστεί το stop the clock έτσι ώστε τουλάχιστον να μην κινδυνέψουμε να χάσουμε τις μικρές ε, επιτυχίες και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αυτή τη στιγμή στον ΙΚΑΟ. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να χάσει και αυτό το μικρό κέρδος που έχουμε σήμερα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να δούμε πού πρέπει να υποχωρήσουμε και αν πρέπει η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποσυρθεί. Δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, επαναλαμβάνω, αυτή η νέα πρόταση. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα σε διεθνές επίπεδο και ότι μπορούν οι τρίτες χώρες να αγνοήσουν και να εμποδίσουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ, κύριε Κόρολα. Thank Είμαι η συγγήτρια της ε, γνωμοδότησης της Επιτροπής Ήτρε. Θα στηρίξω τους Κάλαναν, Κράμερ και Ντέβις. Ε, ελπίζω η υποστήριξη με αυτή να μην υποσκάψει την αξιοπιστία τους. Οι, αλλά, εποχές αλλάζουν. Η στήριξη που είχαν οι αερομεταφορές ε, δεν, την προηγούμενη δεκαετία δεν υφίσταται πλέον, το βλέπουμε αυτό. Και βλέπουμε και τις επιπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο η ιδέα της Κομισιόν δεν πρόκειται να ευοδοθεί. Τα κράτη-μέλη δεν τη στηρίζουν Δεν θέλω να αποτρέψω την Ευρωπαϊκή Ένωση από το να χρησιμοποιήσει ένα εσωτερικό σύστημα ε, ε, εμπορίας ε, δικαιωμάτων. Έτσι κι αλλιώς οι οικονομικές επιπτώσεις είναι μικρές, αλλά οι πολιτικές επιπτώσεις είναι τεράστιες. Η ιδέα της Κομισιόν του να καλύψουμε και τρίτες χώρες με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων είναι παράλογη θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, εμπορικούς πολέμους. Αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Και θα επηρεάσει και την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Ενδεχομένως θα μειώσει και τις επιχειρηματικέ ευκαιρίες και θα πλήξει και τους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς. Το προτινόμενο μοντέλο που ε, ε, θα καλύψει, θα αυξήσει την κάλυψη από το 9 στο 13% των ε, αεροπορικών ταξιδιών. Ακόμα και το περιορισμένο δηλαδή και η περιορισμένη ε, πρόταση ε, δημιουργεί ε, πολιτικά προβλήματα χωρίς να λύνει κάποια περιβαλλοντικά προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι και πάλι έχουμε ένα παράδειγμα για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τέτοια μονομανία με, τα δικά, με το δικό της σύστημα που δεν βλέπει ε, τι προκαλεί αυτό σε άλλους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους. Ε, πολλοί εμπλεκόμενοι λένε ότι ε, Ε, δεν έχουν πρόβλημα στον, το να συμμετέχουν σε ένα σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών, αλλά γιατί θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας το επιβάλλει. Τι είναι αυτό τώρα. Ε, είναι μια πολιτική υπεροψία, ματαιοδοξία. <clears throat> Για όλους αυτούς τους λόγους στην γνωμοδότησή μου στις ΙΤΡΕ θα προτείνω να συνεχίσουμε το σύστημα Stop the Clock ε, ως εσωτερικό ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ε, δικαιωμάτων μέχρι το 2016 και να μην το επιβάλλουμε στους διεθνείς μας εταίρους. Ε, να περιμένουμε την Γενική Συνέλευση του ΙΚΑΟ το 2016 όπου αναμένουμε συνολική συμφωνία Νομίζω ότι για να εξασφαλίσουμε τέτοιου διεθνή συμφωνία θα έπρεπε ε, να ακολουθήσουμε ε, αυτή τη μετριοπαθή στάση ε, και νομίζω θα πετύχουμε τα ίδια αποτελέσματα αλλά με πιο ευφύ τρόπο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κόρολα. Και έχουμε και μία ομάδα επισκεπτών από τη Φιλανδία προσκεκλημένη της κυρίας Κόρολα, τους οποίους χαιρετίζω. Και βεβαίως συνεχίζουμε με τον Μπας Χάσχαλτ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, Ματίας. Υπάρχουν κάποιοι, ότι μισούν, κάποιοι που μισούν το ε, σύστημα εμπορία δικαιωμάτων, το ξέραμε. Ε, αλλά δεν ξέρω. Ε, αν εσύ συμφωνείς Μάρτιν, με τον Κρίς, δεν ξέρω ποιανού η αξιοπιστία πλήττεται περισσότερο. Ε, θα έπρεπε να ανησυχήσει λίγο. Γιατί αν ο Μάρτιν και ο Κρίς αρχίζουν να συμφωνούν, κάτι δεν πάει καλά. Και πράγματι κάτι δεν πάει καλά με αυτή τη συζήτηση. Γιατί ας δούμε από πού ερχόμαστε. Όλοι ξέρουμε ότι ε, οι, οι, οι μεταφορές δεν πληρώνουν τίποτα, παρόλο που η αρχή είναι ο πληρώνει. Όλοι δουλεύουμε για τα συμφέροντα ε, ε, των αεροπορικών εταιριών, των αερομεταφορέων. Ας δούμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε αυτό το σύστημα για τις αερομεταφορές. Γιατί θέλαμε να ε, επιβάλλουμε κάποια, κάποιο σύστημα για τις ε, τιμέ, εκτό και αν ε, καταφέρναμε μια συμφωνία σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό θέλαμε. Διεθνή συμφωνία. Αλλά αν δούμε τη συμφωνία του ΙΚΑΟ, πρώτον, έχουν στόχο για μετά το 2020. Γίνεται δυνατόν ο ένας κλάδος να θέτει το δικό του στόχο. Όλοι οι άδειλοι κλάδοι ζηλεύουν την, αερο, ε, την αεροπορική βιομηχανία. Ε, και μάλιστα λένε ότι μπορούμε ε, ενδεχομένως πριν το 2020 θα αναθεωρήσουν το στόχο τους. Δηλαδή αν το 2009 δεν προλαβαίνουν, μπορεί ο ίδιος ο κλάδο να πει εντάξει, στόχος για αργότερα». Και μετά λένε ότι ενδεχομένως θα καταφέρουν μια συμφωνία 2016, ίσως, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι ήδη ακόμα και σε αυτή τη διεθνή συμφωνία υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις. Το οποίο σημαίνει ότι θα είναι τρίπιο τυρί, γραβιέρα, γεμάτο τρύπες. Αν κάποιοι λένε ότι ο, ο ΙΚΑΟ τα καταφέρει στη Διεθνή Συμφωνία, ξαναδιαβάζουν τη συμφωνία για να δουν τι παραθυράκια έχει. Τώρα, ο Κρίς και ο Μαρτίν ανησυχούν για τη μη συμμόρφωση. Εγώ ανησυχώ για την απουσία πολιτικής βούλησης και όσο λιγότερη πολιτική βούληση έχουμε, τόσο περισσότερη βέβαια έλλειψη συμμόρφωσης θα εμφανίζεται. Βλέπω σε Κρίσ, Κρίς, εσύ πολιτικός όμως και θέτεις ερωτήματα. <laughs> Υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτό είναι ερώτηση που πρέπει να απαντήσει εσύ ο ίδιος. Εσύ έχεις πολιτική βούληση, εσύ Μάρτιν, έχεις πολιτική βούληση, έχεις πολιτική αποφασιστικότητα. Αυτή είναι η ερώτηση. Η πολιτική μας βούληση αμφισβητείται. Και αυτό το βλέπουν στο εξωτερικό, το βλέπουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό έχουμε χάσει αξιοπιστία. Εμείς λέμε θα κάνουμε αυτό αν δεν, έχουν, αν δεν εξασφαλιστεί διεθνή συμφωνία. Και τι κάνουμε, κάνουμε ε, ε, και παρόλο που δεν υπάρχει διεθνή συμφωνία, δεν έχει εξασφαλιστεί, ε, σταματάμε το ρολόι. Και μετά τι κάνουμε, λέμε παρόλο που δεν υπάρχει διεθνή συμφωνία, ας περιορίσουμε την κάλυψη στο δικό μας ε, ενέργειο χώρα και να συνεχίσουμε και το stop the clock. Ε, αυτό υποσκάπτει την αξιοπιστία μας. Γιατί δείχνει ότι δεν έχουμε πολιτική βούληση. Αυτό είναι μια ερώτηση που θα πρέπει να απαντήσουν οι πολιτικοί που είναι εδώ μέσα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο οι αεροπορικές εταιρείες, οι αερομεταφορείς, ακούγοντας τους συντηρητικούς, ακούγοντας τους φιλελεύθερους, θα καταλάβουν ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Συνεπώς, γιατί να μην πολεμήσουν ακόμα πιο ε, σκληρά. Οπότε το θέμα δεν είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση, το θέμα είναι αν εμείς έχουμε την πολιτική βούληση. Οπότε, Πίτερ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που προσπαθείς να κάνεις κάτι, αλλά αυτό που βλέπω εγώ στο κείμενο δεν είναι αρκετό. Αντιπροσωπεύει ήδη μια υποχώρηση λόγω των πιέσεων. Δεν υπάρχει διεθνή συμφωνία. Υπάρχει κάποια κινητικότητα, αλλά δεν υπάρχει διεθνή συμφωνία. Και αν ακολουθήσουμε το δρόμο του, Λί, του Πίτερ Λίζε ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα υποσκάψουμε ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία μας. Για το να προτείνουμε την ε, συνέχιση του Stop the Clock ε, πραγματικά μας γελιοποιεί. Το θέμα είναι αν εμείς έχουμε πολιτική βούληση γιατί δική μας είναι η ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Μπράντι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Όλη αυτή η υπόθεση των εκπομπών και των αεροπορικών εταιριών είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό από όσο φαίνεται γιατί εδώ πέρα φαίνεται το ότι δεν υπάρχει βούληση ή ικανότητα κάτι να κάνουμε για την κλιματική αλλαγή. Να δούμε την αλήθεια κατά πρόσωπα. Δεν έχουμε ούτε ένα, ούτε ένα επιχείρημα που να μας οδηγήσει στο να αδρανίσουμε για τις ε, εκπομπές, τις βλαπτικές των αερομεταφορέων. Και σε αυτό συμφωνούμε. Συνήθως λέμε ότι είναι θέμα οικονομικό. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει οικονομικό θέμα. κοστίζει το, το, το, το επιπλέον πρέπει να πληρωθεί λιγότερο από το καφεδάκι που είναι πριν μπει στο αεροπλάνο. Τα είπε ο Πίτερ Λίζε. Αλλά έχουμε και το θέμα του τι θα γίνει με την ε, τερατώδη αύξηση των εκπομπών στο μέλλον. Είδατε την προβολή, τη στατιστική. Επομένω, δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα, καμιά δικαιολογία για να δρανίσουμε. Ίσιο δίκαιο ανταγωνισμού, εξορισμού, θα είναι έτσι. Υπάρχει εξορισμού. Στο ίδιο ύψος πετούν ε, όλα τα αεροπλάνα. Δεν υπάρχει λόγος, καμία δικαιολογία να δρανίσουμε ούτε σε αυτό το επίπεδο. Και δε, κανείς δεν βιάστηκε να αποφασίσει. Δεν έγινε αυτό από το βράδυ στο πρωί. Το 2008 συζητιέται το πώς θα ενταχθούν στο ΣΕΔΕ οι αεροπορικές εταιρείες. Είπα ναι στην αναβολή πέρσι γιατί θεώρησα ότι είναι βάσιμο το να μην πιέσουμε την ΙΚΑΟ, να μην αποσπάσουμε την, ε, την συμφωνία, αλλά τα ήξερε η ΙΚΑΟ. Ήξερε πού θα κατέληγε το πράγμα εάν δεν υπήρχε συμφωνία. Γι' αυτό και δεν συμφώνησαν. Τίποτα εντυπωσιακό δεν αποφασίστηκε τα είπε και ο συνάδελφος πριν. Νομίζω η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το δικό μας ενεργοχώρο είναι έξυπνη πρόταση. Είναι κάτι πολύ πιο περιορισμένο από την αρχή πρόταση. Αλλά νομίζω θα βοηθήσει να προχωρήσει η υπόθεση που έχει αναλάβει ο Πίτερ Λίζε. Οπότε αφού το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό, τότε τι είναι. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Και αφού είναι μόνο πολιτικό, ε, τότε ας δείξουμε ότι είμαστε μια δύναμη πολιτική που θα πρέπει να σέβονται και να αναγνωρίζουν και οι άλλοι. Αλλά βέβαια αυτό να μην ισχύει μόνο για τα κλιματολογικά, αυτό να ισχύει κάθε φορά που δρούμε ενωμένοι και με αποφασιστικότητα. Γι' αυτό και με ανησυχεί αυτό που συζητούμε σήμερα γιατί δεν πολύ βλέπω ούτε ενιαία στάση, ούτε αποφασιστικό του Πλευράς Κοινοβουλίου. Εάν δράσουμε δυναμικά, τότε θα δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε πρωτοπόροι για τα θέματα του περιβάλλοντος και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Οπότε ευχαριστούμε στην για την έκθεσή σου και ελπίζω να εγκριθεί ταχαίως. Ευχαριστώ κύριο Ζέμπερ. Ευχαριστώ. Εγώ στηρίζω την πρόταση του εισηγητή, του Πετερλίζε και νομίζω ότι από νομικής απόψεως, όπως έδειξε η μέχρι τώρα συζήτηση, δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης. Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν ναι ή όχι λαμβάνουμε τον εαυτό μας τα σοβαρά. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά παίρνει αποφάσεις ε, μόνη της, ανεξάρτητα ή αν κάποιοι μας επιβάλλουν πιέσεις ε, και αποφάσεις. Αν τα κράτη-μέλη είναι κυρίαρχα και μπορούν να αποφασίσουν, γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα συνεχίζουν να παίζουν το ίδιο στρατηγικό παλιό παιχνίδι και το σημαντικό πρόβλημα βεβαίως δεν είναι το ύψος των τελών. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ παίρνει μια ενιαία θέση, μια τοποθέτηση όπως είπε και ο Πίτερ Λίζε και μπορεί να βαρύνει, να επιβάλλει κάτι. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Αυτή είναι η ουσία. Θέλουμε να δράσουμε από κοινού. Επαναλαμβάνω δεν υπάρχει νομικό θέμα. Από νομικής απόψεως κανείς δεν αμφισβητεί την απόφαση αυτή ή θέλουμε να μας επιβάλλει κάποιος άλλος από τα έξω μία απόφαση. Θέλουμε να γελιοποιηθούμε διεθνώς. Γιατί αυτά είναι μέτρα που πραγματικά καλούμεθα να αποφασίσουμε ανεξάρτητα. Και εδώ έχουμε μία δυνατότητα να το κάνουμε. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Αλλά μέχρι τώρα στην, ε, στην ιστορία, σαφώς και έχουμε και, και από άλλες περιπτώσεις, και εγώ έχω και από τη δική μου προσωπική ιστορία, ε, πολλές ευκαιρίες που μας δείχνουν ότι μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι από τη στιγμή που είμαστε ενωμένοι. Εδώ έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα, γιατί δεν είμαστε αρκετά ισχυροί η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύστημα, σαν ενέργειος χώρος ε, έχει την βαρύτητα που έχει. Το θέμα είναι όμως ότι η αξιοπιστία μας θα πληγεί και δεν υπάρχει περίπτωση να μας πάρει κανείς σοβαρά εάν δεν μπορούμε σε ένα τέτοιο θέμα να επιβάλλουμε τα επιχείρηματά μας. Εδώ μιλάμε για εμπορικούς πολέμους, για μεγάλες διαμάχες και διενέξεις στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών. Δεν πρόκειται για κάτι τόσο μεγάλο επίβολο. Ελπίζω όμως, ελπίζω, όπως είπε και ο Πίτερ Λίζε, να πάρουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας και ελπίζω να κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα που να είναι ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα αποφασίσουν κάτι που να έχει επίπτωση στον προϋπολογισμό. Θα πάρουμε επιτέλους μια κοινή απόφαση που αφορά τα οικονομικά, τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πρόκληση. Ας μην υποχωρήσουμε πριν το δοκιμάσουμε. Ε, μακροπρόθεσμα έχει νόημα αυτό που κάνουμε. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν πρέπει να υποχωρήσουμε. Ας πάρουμε μια κυρία απόφαση, γιατί μακροπρόθεσμα μόνο αυτό είναι πρόοδος. Εάν δεν προχωρήσουμε ομόφωνα πραγματικά είναι πολύ κρίμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, ευχαριστώ, Ρίχα Τσέμπερ. Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση εδώ δεν μπορούμε από εθνικής απόψεως να πούμε ότι όλοι έχουν κοινέ θέσεις, αλλά κάπως έτσι παρουσιάζεται. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάθε πρωί περπατάω μέχρι εδώ Και όταν υπάρχει ομίχλη και σύννεφα, λίγες μέρες το χρόνο δηλαδή, βλέπει κανείς νωρίς το πρωί σε 7.30 τον ουρανό γεμάτο από ίχνη εκπομπών αεροπλάνων. Γεμάτο. Κάθε πρωί. Και αυτό είναι σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε. Η ενέργεια κυκλοφορία αυξάνεται πολύ γρήγορα. Και εμείς ως πολιτικοί όλοι μας θα πρέπει να το σκεφτούμε. Να σκεφτούμε το περιβάλλον. Να σκεφτούμε τη μελλοντική ζωή, τη ζωή των παιδιών μας. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι θέμα συνείδησης. Πώς θα ζούμε μετά από 10-20 χρόνια αν δεν αλλάξουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε κάποιες λύσεις. Χρειαζόμαστε κάποια αλλαγή. Δεν είναι όλες οι λύσεις σωστές, αλλά χρειαζόμαστε κάποια αλλαγή και χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η κατάσταση και πού βαίνουμε τι συμβαίνει πάνω από τα κεφάλια μας. Ίσως οι άνθρωποι που ζουν στις μεγάλες πόλεις δεν αντιδρούν και εγώ αντιδρώ γιατί έρχομαι από μια χώρα που δεν είναι τόσο μολυσμένη. δεν θα επικρίνω τις ε, προτάσεις της Κομισιόν. Ε, πρέπει να βρούμε μία λύση. Ο καθένας μας ας συνεισφέρει αυτό που επιθυμεί, αλλά μία λύση πρέπει να τη βρούμε. Ας προτείνουμε βελτιώσεις. Δεν μπορούμε όμως να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Ας σκεφτούμε και την τεχνολογία τι τεχνολογία χρειάζεται. Γιατί με αυτό το ρυθμό μετά από 30-40 χρόνια δεν θα μπορούμε να ζούμε όπως ζούμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, εδώ είναι ο ενέριο χώρος. 2.000 πτήσεις έχουμε σε όλο τον αέριο χώρο. Κυρία Κόρολα. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Θα ήθελα να πω ότι αυτοί τους που έχουν προσκαλέσει είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων και ε, είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων στη χαλιβουργία και δυστυχώ κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι είναι ε, αστείο. Εγώ ανησυχώ για την ε, απασχόληση στην Ευρώπη γιατί όσον αφορά τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε και τι εκπομπέ είναι μια χαρά η Χαλιβουργία στην ε, Φινλανδία. Οπότε γι' αυτό και προβληματίζομαι που ε, ε, έτσι, έτσι όπως έχει σήμερα το κλίμα στην απασχόληση ουσιαστικά παροξύνουμε την ανεργία. Ο πρόεδρος. Κάτι δεν κατάλαβα καλά. Μιλήσατε για τη χαλιβουργία. Και εμείς έχουμε αυτή τη δραστηριότητα στη δική μου επικράτεια, στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Και εμείς έχουμε χαλιβουργία και καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι, βεβαίως ε, το θέμα αυτό μας απασχολεί όλους, το θέμα της απασχόλησης. Θα δώσω τώρα όμως το λόγο στην Επιτροπή. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο να απαντήσετε σε κάποια σημεία και κατόπιν θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους αξιότιμους βουλευτές για όλη αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που σίγουρα πρέπει να μας βοηθήσει στον προβληματισμό μας. Είναι η κατάσταση περίπλοκη πολιτικά. Είναι μια μεγάλη πρόκληση και απαιτεί υπεύθυνη αντιμετώπιση από όλους τους εμπλεκομένους. Και βέβαια θα είναι σημαντικό το να αντιδράσουμε ταχαίως, να έχουμε μέχρι το τέλος του Απριλίου νομική βάση και θα πρέπει μέσα επικοδομητικά να ασχοληθούμε όλοι, όλοι, όλοι αυτοί που θα συμμετάσχουμε στην ε, συναπόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε θεώρησε ότι η δράση η σφαιρική, η παγκόσμια, η ολοκληρωμένη είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις δραστηριότητες και γι' αυτό και εμείς λέμε, είχαμε πει πέρσι να ε, κάνουμε αυτή την ε, αυτό το, το διάλειμμα ας πούμε, όχι για λόγους αδράνειας, αλλά για να δούμε τι, θα, τι θέλουν οι τρίτες χώρες, οι εταίροι μας, να δούμε πώς βλέπουν αυτά τα πράγματα, να αναζητήσουμε κάποιες λύσεις ε, θετικές και συναντικές και κάτι το οποίο μας είπαν ότι προτιμούν είναι να έχουμε μία προσέγγιση ε, που να έχει σχέση, σαν να έχει σαν κριτήριο τον εναέριο χώρο και έγιναν κάποια πράγματα πρόοδο στην συνέλευση του ΙΚΑΟ που ήταν πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Οπότε εμεί συνεχίζουμε να θέλουμε την επιτυχία των προτάσεών μας. Είπα κάποιοι βουλευτές ότι δεν ήταν τόσο σωστό του να κάνουμε πίσω σε σχέση με που είχαμε στην αρχή προτείνει, αλλά δεν είναι έτσι. Θα πρέπει μέχρι το 2020 να περιμένουμε να δούμε τι ισχύει και να δούμε μετά τι μέτρα θα προτείνουμε. Οπότε θα πρέπει γι' αυτό να δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσουμε τα όσα θέλουμε να την πλευρά περιβάλλοντος και στις νέες μεταφορές. Για μας είναι πάρα πολύ ψηλή προτεραιότητα. Και για την ισοδαφικότητα, όπως ζήτησαν οι εταίροι μας, οι τρίτες χώρες, είπαμε ότι αυτό είναι κάτι το θεμητό και γι' αυτό και τελικά είχαμε θετική εξέλιξη των επαφών και διαπραγματεύσεων. Να μην υπάρχουν δυσμενείς διακρίσεις, και υπάρχουν ισχυροί ανταγωνισμού σχέση με τα δρομολόγια των αερομεταφοριών. Θεωρούμε ότι κάναμε ό,τι παίρνει από το χέρι μα, ώστε να ε, ενεργήσουμε στο πνεύμα των αποφάσεων η ΚΑΟ. Υπάρχουν κάποιε διατάξει στο κείμενό μα που ακριβώ απηχούν τι απόψει τη ΚΑΟ, όμω παρόλα αυτά επιφυλαχθήκαμε όσον αφορά κάποια τα οποία είπε η ΚΑΟ, αλλά θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ότι εμείς για να λάβουμε δράση θα έπρεπε να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη ε, κάποιων κρατών, κάποιων αερομεταφορέων που επιχειρούν στην Ευρώπη. Αν κάποιος ε, έχει εμπορική δράση παγκόσμια, κάθε φορά θα πρέπει να σέβεται το δίκαιο του χώρου όπου ενεργεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να τηρηθεί το κοινωτικό δίκαιο. Έριξα μια ματιά στις ε, τροπολογίες του κ. Λίζε. Δεν καλύφθηκαν από τη δική μας πρόταση και αυτό γιατί θέλαμε να ενεργήσουμε ταχαίως με σύντομο κείμενο γιατί αν, έχουμε, αν αρχίσουμε τώρα ε, τι τις εκβάθρων αλλαγές στο κειμένο είπαμε ότι θα περιπλακεί η διαδικασία στην απόφαση και γι' αυτό και ελαχιστοποίησαμε τις ε, αλλαγές που κάναμε. Όμως, από την άλλη μεριά, είπαμε ότι θέλουμε οπωσδήποτε οι επιπτώσεις περιβαλλοντικές να είναι σίγουρες αυτές που θέλουμε. Και συμφωνώ 100% με μια σειρά βουλευτών που είπαν ότι η εφαρμογή είναι προϋπόθεση αξιοπιστίας της ε, πολιτικής ε, της Ένωσης το 2012 που σταματήσαμε και περιμένουμε θα πούνε οι εταίροι είπαμε ότι καλύπτεται των... Είχαμε, είχα, είχαμε συμμόρφωση 2012 και από τους Ρώσους και από, και από άλλους. Όλων όσους είχαν τότε εμπλακεί ε, σε συνομιλίες και διαπραγματεύσεις. Είναι σαφές ότι υπάρχει οφαστικότητα, υπάρχει η βούληση. Να δούμε το πώς ε, το ΣΕΔΕ στο μέλλον θα γίνει σεβαστό, θα εφαρμοστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πρέπει να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί στηρίζει την πρότασή μας. Νομίζω ότι έτσι οι προτάσεις μας πρόκειται να προχωρήσουν, να ευδοκιμήσουν και να εφαρμοστούν. Εμείς με όλους τους εταίρους μας θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια διαδικασία, στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματο, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέχρι τα τέλη Απριλίου, όπω προβλέπετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, για να ολοκληρώσει, ο εισηγητή έχει το λόγο, Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχήν όλους όσους στηρίζουν την πρότασή μου. Είναι κρίμα που αυτό δεν το κάνουν όλοι αλλά εν πάση περιπτώσει άκουσα πολύ προσεκτικά αυτούς που επικρίνουν το κείμενό μου. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξο, κάποιοι το θεωρούν πολύ φιλόδοξο. Ίσως θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε λοιπόν κάπου στη μέση, σε μια πρόταση πιο μετριοπαθή. Εγώ πάντως ε, άκουσα πολύ προσεκτικά τους μεν και τους δε και θεωρώ ότι είναι η πρότασή μου ήδη στο μέσο μεταξύ δηλαδή των δύο ακραίων ε, προτάσεων. Άκουσα τους πράσινους, την Αχάση που προτείνουν να επεκταθεί η πρόταση. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε και ακούγοντας αυτούς που είναι αντίθετοι να προτείνουμε κάτι τέτοιο. Από άποψη περιβαλλοντοϊκής ναι, Μπορούμε να το κάνουμε. Από άποψη νομική επίση, Αλλά σήμερα βλέπουμε το, τον ΙΚΑΟ να κάνει μια μικρή κίνηση προς την πρότασή μας. Ας παραμείνουμε λοιπόν σε αυτό και ας μην ε, χάσουμε και τα λίγα που έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυτά που ακούω πολλές φορές με ξαφνιάζουν. Η η Ντάκμα Ροντμπέρεντ όσον αφορά άλλα θέματα όπως την φαρμακοεπαγρύπνηση παραδείγματο χάρη βλέπουμε να ακούγονται πολύ φιλόδοξες και ακραίες τοποθετήσεις της συζήτησης στην Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια όλα αυτά ξεφουσκώνουν. Θα πρέπει να, στην προκειμένη περίπτωση να δώσουμε εντολή και αυτό πρέπει να γίνει πριν τις 30 Ιανουαρίου. Εγώ πραγματικά ξαφνιάστηκα ακούγοντας ε, συναδέλφους όπως την Ρίτα Κόρολα που λένε ότι εντάξει μπορούμε να το δεχθούμε. Ας είμαστε συγκεκριμένοι. Εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξέρουμε αν ναι ή όχι πρόκειται για στρέβλωση του ανταγωνισμού και αν πραγματικά επιβαρύνουμε υπερβολικά τις αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης. Είναι χαμηλό αυτό που προσπαθούμε να επιβάλλουμε ή δεν είναι χαμηλό. Τους επιβαρύνουμε ή δεν τους επιβαρύνουμε. Υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ναι ή όχι. Και εγώ πήρα επιστολές πολύ αγριεμένες από πολλούς όταν δεχτήκαμε την πάυση, το stop the clock. Και κάποιοι που θυμούνται τι είχαμε αποφασίσει πριν από μερικά χρόνια, σίγουρα ε, δεν μπορούν να γνωρίσουν ότι όταν δεχτήκαμε αυτήν την πάυση, αυτήν την, αυτό το stop the clock, το δεχτήκαμε για ένα χρόνο. Αυτός ο χρόνος λύγει. Αν λοιπόν δεν ε, λάβουμε υπόψη μας το τι συμβαίνει διεθνώς, όντως θα καταντήσει η ευρωπαϊκή, ο ευρωπαϊκός τομέας των αεροπορικών ε, μεταφορών να υποστεί πλήγμα. Γι' αυτό και προσπαθούμε να μην δημιουργήσουμε μειονεκτικές συνθήκες για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Επαναλαμβάνω, αποφασίστε είναι ή δεν είναι στρέβλωση ανταγωνισμού, είναι ή δεν είναι επιβάρυνση. Για μένα είναι δύσκολο να ε, πηγαίνουμε ένα βήμα αριστερά και ένα βήμα δεξιά. Άκουσα πολύ προσεκτικά επίσης και αυτού σαν τον ε, Chris Davis, το θέμα της συμμόρφωσης. Ναι, το θέμα της συμμόρφωσης με το stop the clock δημιουργεί πρόβλημα, γιατί σήμερα υπάρχουν ε, κράτη-μέλη που δεν λαμβάνουν υπόψη τους το σύστημα της αεροπορικές εταιρείε της ε, Κίνας ή της ε, Ινδίας. Υπάρχει λοιπόν συμμόρφωση ή δεν υπάρχει. Εδώ συζητούμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι οι περισσότεροι ακολουθούν το σύστημα. Υπάρχουν και κάποιοι αερομεταφορείς οι οποίοι για την εικόνα τους, ε, για λόγους διαφήμισης, ενώ δεν είναι υποχρεωμένοι, το κάνουν. Συμμορφώνονται. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν πρόβλημα με την νέα αυτή πρόταση, Μάρτιν και υποστήριξαν την πρόταση αυτή στον ΙΚΑΟ. Και τι να σας πω, στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπως ξέρετε, είναι ιερός ο Αμερικανικός εναέριος χώρος. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί είναι ιερές. Και σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι κάτι που αποφασίστηκε δεν θα το τηρήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινέ προκλήσεις με τους Αμερικανούς και κάθε φορά που αποφασίζουμε ένα νομικό κείμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να κοιτάμε το θέμα της υλοποίησης, της εφαρμογής. Εγώ στη δική μου εκλογική περιφέρεια έχω επαφές με επιχειρηματίες και εγώ έχω στη Γερμανία βιομήχανους στον τομέα του, της χαλιβουργίας, δεν είναι μόνο στη Φιλανδία, οι υπερσύγχρονες χαλιβουργίες και στη Γερμανία έχουμε. Και σίγουρα υπάρχει βελτίωση που μπορεί να γίνει, αλλά αν συγκρίνουμε την κατάσταση στην Κίνα με την Ιταλία ή τη Γαλλία, καταλαβαίνετε ότι ο τομέας της χαλιβουργίας στην Κίνα λειτουργεί με συστήματα και την ίδια, τα οποία δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά στάνταρτς και βεβαίως την ίδια ώρα οι Κινέζοι μας εμποδίζουν να νομοθετήσουμε στον τομέα των αερομεταφορών. Τι θα πει η κυρία Κόρολα και ο Μάρτιν Κέλεμαν όταν επικαλεστούμε αυτά τα επιχειρήματα. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να πάρουμε μια απόφαση για μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, ένα νομοθετικό κείμενο, τον οποίο θα επιβάλλουμε και θα εφαρμόσουμε στην Ευρώπη επειδή μας πιέζουν άνθρωποι, χώρες που έχουν άλλα πρότυπα, άλλη νομοθεσία και κατόπιν ανταγωνίζονται και μας πιέζουν κιόλας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών, ξεκίνησε αυτές τις διαπραγματεύσεις το 2008. Το Συμβούλιο το ξεκίνησε αυτό. Ήταν πρωτοβουλία του Συμβουλίου. Δεν ήταν ούτε του Κοινοβουλίου ούτε της Επιτροπής. Και η απόφαση που ελήφθη τότε να συμπεριληφθεί ο εναέριος χώρος στο σύστημα εμπορίας εκπομπών απλώς δεν εφαρμόστηκε. Και αυτό λέμε να κάνουμε σήμερα. Ας αφήσουμε λοιπόν τις πιέσεις και τις απειλές. Υπάρχουν απειλές. Αλλά αν υπάρχει νομοθεσία, θα πρέπει να την εφαρμόσουμε, να την τηρήσουμε. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν, νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η αδυναμία είναι βεβαίως ότι δεν ξέρουμε πόσο θα χρησιμοποιηθούν από εδώ και πέρα οι νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να μην ε, επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο το περιβάλλον, να μειώσουμε τις ε, συνέπειες ε, στις αλλαγές του κλίματος. Είναι θέμα και οικονομικό αλλά κυρίως αποτελεσματικότητας. Τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο ε, θέμα εδώ, να δεχτούν το σκοπό αυτής της προσπάθειας. δεν είναι βέβαια ο μόνος τομέας, δεν είναι μόνο νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα, ένα θέμα αρχής και θα πρέπει να σταματήσουμε να απορρίπτουμε αυτές ε, τις προτάσεις για υποχώρηση συμβιβαστικής προτάσεις πιο αδύναμες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Πίτερ Λίζε. 19 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι. Θα συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή της Τροπολογίας στις 20 ε, Ιανουαρίου. Θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή στις 30 Ιανουαρίου. Και προβλέπεται να συζητηθεί τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με το σημείο αυτό. Μπορούμε να περάσουμε στο 23 που είναι η ανταλλαγή απόψεων με την ΑΤ με την ασφάλεια της ανθρώπινης κατανάλωσης της ασπαρτάμης. Θα δώσω το λόγο αμέσως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Σας παρακαλώ, αν δεν θέλετε να συζητήσετε το θέμα αυτό. Μπορείτε να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Διακόψτε μου για ένα λεπτό. So, ich glaube, jetzt können Sie starten. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Έχετε το λόγο. Uh, thank you, Chair. Uh, my name... Γεια σας. Με συνοδεύουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν τεχνικές γνώσεις για το θέμα το οποίο συζητούμε. Αν συμφωνείτε, θα πρότεινα ε, να κάνουμε μια εισαγωγή τριών ως πέντε λεπτών για το θέμα. Συμφωνείτε? Ωραία. Να πω λοιπόν καταρχήν ότι είναι το, η πρώτη γλυκαντική ουσία η οποία αξιολογείται σε ένα πρόγραμμα το οποίο λύγει το 2020. Η αρχή της ε, επαναξιολόγησης των γλυκανικών ουσιών είναι ότι αυτή τη φορά όλες οι πληροφορίες συλλέγονται από την ΕΦΣΑ. Ε, δεν υποβάλλονται από κανέναν. Ε, χρησιμοποίησαμε βέβαια μια, τις δικές μας ερεύνες αλλά και καλέσαμε ε, όλους, όσους έχουν τέτοιου πληροφορίες να τις καταθέσουν. Ε, δημιουργήσαμε ένα πάνελ το οποίο ε, έλαβε όλες τις ε, πληροφορίες και έκανε μια πλήρη τοξικολογική μελέτη. Θα δώσω το λόγο στους αδέλφους μου, τον συνάδελφο κύριο Κάς, δόκτωρα Κάς, αλλά να σας πω ότι προεπήμεν και σε δημόσια διαβούλευση, μέσω της οποίας πήραμε πολύ input. Ήταν πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες οι οποίες μας δόθηκαν μέσω της δημόσιας διαβούλευσης και που επηρέασαν ε, την, το προσχέδιο γνωμοδότησής μας. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν να δώσω το λόγο στον Δόκτρα Κάς, ο οποίος θα σας παρουσιάσει τα επιστημονικά πορίσματα. Ευχαριστώ. Πρώτο σημείο, σε ό,τι αφορά την ε, χημική δομή της ασπαρτάμης. Είναι ένα απλό μόριο δύο βασικές μονάδες, πρωτεϊνικές μονάδες, αμινοξέα μάλλον. Φιναλίνη και ασπαρτικόξι. Ε, τροποποιείται χημικά για να τους δώσουμε την γλυκή, τη γλυκιά της γεύση. Ε, στον οργανισμό ε, αποδομείται και παράγει μεθανόλη, ασπαρταμικό οξύ κλπ. κλπ. Αλλά δεν φτάνει ποτέ ως ασπαρτάμι στα όργανά μας, δεν μπαίνει ποτέ ε, ως ασπαρτάμι στο αίμα. Ε, δημιουργούνται αμινοξέα, όπως οποιαδήποτε αμινοξέα παίρνετε μέσω του πρωινού σας για παράδειγμα. Ε, τι γίνεται όμως με τη μεθανόλη. Η μεθανόλη είναι ιδιαίτερη η περίπτωση. Η μεθανόλη είναι ίδια με την μεθανόλη η οποία κλείεται από ε, τις των προκυπευτικών που τρώμε. Η μεθανόλη παράγεται και με φυσικό τρόπο και σε μεγάλες ποσότητες από το σώμα μας γιατί χρειάζεται σε πολλές χημικές αντιδράσεις στα όργανά μας και στα κύτταρά μας. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πλήρως τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, να σας ε, να περιοριστώ στην αξιολόγηση περί ε, τοξικότητας και καρκινογένεσης. Ερώτηση λοιπόν, προκαλεί καρκίνο ασπαρτάμι. Έχουμε οκτώ μελέτες σε ποντίκια. Ε, τα τελευταία 40 χρόνια καμία από αυτές τις μελέτες δεν ε, περιλαμβάνει ενδείξεις ότι η ασπαρτάμι προκαλεί καρκίνο. Όμως γνωρίζουμε και δύο μελέτες ε, που ισχυρίζονται ότι προκαλεί λιφώματα σε ποντίκια. Η ΕΦΣΑ ανέλησε τα στοιχεία και εντόπισε προβλήματα ε, ε, πνευμονολογικά σε τέτοιου ποντίκια. Ε, Αξιολογήσαμε και τις ε, μελέτες που έχουν γίνει, ε, όπως και πήραμε υπόψη και τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει από αμερικανικές, ε, ε, αμερικανικά Ινστιτούτα. Ε, οι πνευμονικές λοιμώξεις ε, ε, είχαν από ό,τι φαίνεται παρερμηνευθεί και είχαν θεωρηθεί λυμφώματα. Δεν ήταν όμως λυμφώματα. παρόμοιες, ε, παρόμοιες, ε, παρόμοια επιχειρήματα και παρόμοιες μελέτες που ε, κατήγγυλαν άλλου τέτοιου τύπου περιστατικά είχαν επίσης εντοπιστεί και είχαν αναλυθεί από εμά και είχαν θεωρηθεί και παλιότερα ως αβάσιμες. Τώρα, τι γίνεται με την εγκυμοσύνη. Ε, οι ψηλές δόσεις ασπαρτάμις είχαν ε, δείξει ε, ε, μικρές ανομαλίες στα έμβρια και μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης, καθώς επίσης και αυξημένη τοξικότητα του στο αίμα. σε, η βασική παρατήρηση ήταν ότι σε πολλές μελέτες η ασπαρτάμι είχε ελεγχθεί μαζί με τους μεταβολιστές της, όπως η φιναλαναλίνη. Η φιναλαναλίνη ε, δημιουργεί τα ίδια αποτελέσματα στα έγκια ποντίκια όπως και η ασπαρτάμι. Αυτό οδήγησε στην υπόθεση ότι η ασπαρτάμι ε, δημιουργεί αυτά τα αποτελέσματα στα έγκια ποντίκια εξαιτία της φιναλαναλίνης. Έχει λογική, γιατί πράγματι είναι ένα τοξικό μηνόξι η φιναλαναλίνη. Η φεναλκετονουρία και για παράδειγμα είναι μια κληρονομική ασθένεια η οποία ε, οφείλεται στην ε, αδυναμία διάσπασης φιναλαναλίνης και αυτό οδηγεί σε υψηλή τοξικότητα ε, ιδιαίτερα σε έγκια ποντίκια. Γνωρίζουμε πολλά για αυτή την ασθένεια και, της ε, και για τη φιναλαναλίνη. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν κλινικές κατευθυντές γραμμές σε όλο τον κόσμο ε, που καθορίζουν ποια ε, ε, είναι η ασφαλής ποσότητα της φιναλαναλίνης στο αίμα. Το πάνελ έκανε και μια μοντελοποίηση για να προβλέψει τα επίπεδα φιναλαναλίνης που θα οφείλονται σε κατανάλωση ασπαρτάμης. Από τους υπολογισμούς μας κατέστησε σαφές ότι η κατανάλωση ακόμα και 40 μιλιγράμμ ε, ασπαρτάμις ανά κιλό βάρους του σώματος δεν θα έδινε φιναλαναλίνη σε περιεκτικότητα στο αίμα τόσο ψηλή όσο να μας ανησυχεί. Θα μπορούσατε μάλιστα να παίρνετε αυτά τα 40 μιλιγκράμμ κάθε ώρα, όχι όλη τη μέρα, και πάλι δεν θα φτάνατε σε αυτό το επίπεδο φιναλαναλίνη στο αίμα. Συνεπώς, τα συμπεράσματα είναι ότι η ασπαρτάμι δεν προκαλεί καρκίνο, ούτε και αποτελεί κίνδυνο για τον αναπτυσσόμενο έμβριο με τις ε, συνιστόμενες ημερήσιες ποσότητες. Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι η είναι ασφαλίζει για ανθρώπινη κατανάλωση και δεν χρειάζεται να αναθεωρηθεί η ημερήσια ε, ε, συνιστόμενη ποσότητα των 40 μιλιγκράμμ αλλά ανά ε, κιλοβάρους. Τέλος, το ερώτημα είναι αν μας εκπλήσει ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας για την ασπαρτάμια αυτή τη στιγμή. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί, Γιατί η ασπαρτάμι από μόνη της δεν μπαίνει στο σώμα. Αποσυντίθεται στα έντερα και ε, παράγει τρία φυσικά προϊόντα, όπως σας είπα. Η αξιολόγησή μας έδειξε ότι η φιναλαλίνη, το ασπαρτικό οξύ και οι μεθανόλοι που παράγονται, ακόμα και στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα αντιπροσωπεύουν το πολύ το 10% ε, των, ε, της ε, ποσότητας που πρέπει να λαμβάνεται από αυτούς τους μεταβολιστές. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ο πρώτος ο οποίος θα λάβει το λόγο. Σύμφωνα με τον κατάλογο των αγοριτών που έχουν εγγραφεί, Πίτερ Λίζε, Λίνε Μακάβαν, κυρία Λεπάζ. Πίτερ Λίζε, πρώτος, συ. Όχι, όχι, Ελίνα μπορεί να λάβει εσύ το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η κυρία Ρότμπερν που έπρεπε να φύγει μου είπε να ρωτήσω κάτι εξ ονόματος. Θέλει να μάθει τι γίνεται όσον αφορά την αντίθεση συμφερόντων, σύγκρουση σύμφωνα για αυτού οι οποίοι τώρα έχουν εμπλακεί στην τα τελευταία πέντε χρόνια. Μπορεί έτσι να μας πει αν κάποιοι εξ αυτών έχουν εργαστεί γιατί στην σχετική βιομηχανία παραγωγής αυτών των γλυκαντικών. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η υπόθεση, λέει κυρία Λεπάζη, για την Εύσα και την Ασπαρτάμι είναι ένα θέμα το οποίο πέρασε από πολλούς, πολλούς μέχρι με έναν εδώ πέρα. Θα πρέπει να κάνουμε αυτή σίγουρα. Και εδώ πέρα πάρα έχουμε καταδείξει ότι αυτές οι μελέτε που ήταν η βάση του προβληματισμού και δόθηκαν η εγκρίση για την κυκλοφορία και θέση που στην αγορά είναι αυτά τα οποία ε, δεν τα έχει βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως μας λέει τώρα και η ΕΦΣΑ. Δεν είχε στα χέρια της, οπότε και τώρα είχαμε ε, τις μελέτες που ξεκίνησαν το 2012 και τα πάντα και το 2020 και είχαμε τώρα αυτές τις πρώτες ε, μελέτες, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο και οπότε ε, άρχισαν τότε ε, οι αμφισβητήσεις κυρίως από πλευράς ε, ε, Ιταλών και Δανών ε, επιστημόνων οι οποίοι κατέδειξαν με κάποιες μελέτες ποιες είναι οι επιπτώσεις, οι συνέπειες της ασπαρτάμης επί του εμβρίου και ποιο είναι το πρόβλημα για τις εγγύους. Ο επίσης ε, κατέδειξαν ότι είχαν απλώς αντιγράψει μια μελή του 2007 από την ομάδα Μπέρντοκ. Σε περίπου 100 γραμμές λοιπόν ξαναλέγαν τα ίδια. Σε αυτή την δίθεν νέα εργασία πάντως τώρα θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την ΕΦΣΑ γιατί έκανε τον κόπο να απαντήσει στις παρατηρήσεις μας μετά από αυτές τις ε, διαβουλεύσεις παρά το ότι σε μερικά σημεία ήταν πολύ λακωνικός η εκπρόσωπη της ΕΦΣΑ Ακούσαμε τι είπε και η κυρία, Εύσα, η κυρία Μακαβάνη και γι' αυτό έχουμε υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι σημαντικό η ΕΦΣΑ εφαρμόζει σύστημα δύο μέτρων και 2 σταθμών. Έχουμε 66 μελέτες που καταδεικνύουν ότι η ασπαρταμ είναι ασφαλής. 53 είναι και 13 δεν είναι αξιόπιστες λέει η ΕΦΣΑ. Έχουμε πολλές μελέτες που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ασπαρτάμι και τίποτα από αυτά δεν τα θεωρεί αξιόπιστα η ΕΦΣΑ. Δεν καταλαβαίνω. Πώς είναι δυνατόν. Όλες οι μελέτες λαμβάνονται υπόψη όταν λένε ότι είναι αξιόπιστοι. Και αυτές που λένε το ανάποδο δεν είναι αξιόπιστες. Ακριβώς όπως έγινε με την... Την πεις φαινόλη. Αυτά είναι παράδεκτα. Το σου το μάλλον καθώς η βάση της μεγής επιτρεπόμενης ημερησίας δόσης σύμφωνα με την ΕΦΣΑ, στηρίζεται σε μελέτες της βιομηχανίας του 1973 που δεν είναι α, επιστημονικές. Συνήθως λαμβάνονται υπόψη επιστημονικές μελέτες. Δεν σχέση αυτό με την ασπαρτάμε. Επίσης, οι περισσότερε από αυτές τις μελέτες που μας λέει το ΕΦΣΑ είναι μελέτε που ποτέ δεν δημοσιεύτηκαν. Δηλαδή υπάρχουν στεγανές βάρο αυτών που αμφισβητούν την ασπαρτάνη. Δεν είναι δυνατόν να μας ικανοποιεί το ότι καμία δυσμενής μελέτη δεν έχει αναδειχθεί. Έχουμε εδώ πέρα ουσιαστικά μόνο τις μελέτες που έχουν χρηματοδοτηθεί από τη βιομηχανία. Επίσης, θα ήθελα να μάθω τι έγινε με εκείνο το εργαστήριο που έκανε κάποιες ε, ε μελέτες που, από αυτό το εργαστήριο που κρίθηκε απαράδεκτο από την ΕΦΣΑ το 1976. Αυτά, Πρόεδρε έχω πάρα πολλές σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την επανεξιολόγηση της ΕΦΣΑ. Αναδύονται ακριβώς τα ίδια ερωτήματα αυτά τα οποία έθεσε και η κυρία Ροτ Μπέρεν, ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κυρία Λεπάζ, Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με τις δύο προηγούμενες συναδέλφους όσον αφορά την ε, επαναξιολόγηση. Θυμάμαι ότι το 2012 ένας ε, επιστήμονας από την ε, ΕΑΤ είχε πει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία καμία απολύτως αμφιβολία και ότι η μελέτη η οποία ουσιαστικά πρόκειται για επαναξιολόγηση, δεν πρόκειται και καινούργια μελέτη σε καμία περίπτωση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την ασπαρτάμι και ότι δεν έχει αρνητικά αποτελέσματα επί της υγείας. Θα ήθελα όμως να μου πείτε πώς είναι δυνατόν επί των 55 μελετών που έχουν γίνει, όλες να μην λαμβάνονται υπόψη καθότι δεν είναι αξιόπιστες. Δηλαδή τίποτα από αυτές τις 55 δεν είναι βάσιμο, κανένα στοιχείο, κανένα συμπέρασμα. Το θεωρώ πολύ παράξενο αυτό. Επίσης υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες για την ασφάλεια των τροφίμων στα κρατημέλη που αντίθετα θεωρούν βάσιμες κάποιες από αυτές τις μελέτες. Όλες αυτές οι αρχές δεν λαμβάνονται υπόψη από τον ε, Οργανισμό Ασφάλισης Τροφίμων στην Ευρώπη. Υπάρχουν επίσης και πάρα πολλά σφάλματα όσον αφορά τις αποδείξεις, λανθασμένα στοιχεία, αβάσιμα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τις ε, μελέτες αυτές, τις οποίες λαμβάνει υπόψη της ΙΑΤ. Ε, Πώς είναι λοιπόν δυνατόν όλα αυτά τα σφάλματα να μην διορθώνονται. Η μελέτη της ΕΑΤ έτσι και αλλιώς μας δείχνει ότι εδώ λαμβάνονται υπόψη δύο μέτρα και δύο σταθμά και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ασπαρτάμι δεν είναι βλαβερή χρησιμοποιώντας εντελώς παράξενες διαδικασίες. Δεν είμαι καθόλου ήσυχη και δεν είμαι η μόνη και νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και με τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε 1,5 λεπτό κύριε Γιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για ένα σκάνδαλο και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Καθότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων χρησιμοποιεί αβάσιμα στοιχεία και αυτό το λέω και προς τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και προς ε, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλής Τροφίμων. Είναι θέμα δεοντολογίας και πρέπει να πούμε πολύ ξεκάθαρα εμείς οι Ευρωπαίοι Ευρωβουλευτές θέλουμε να ασκήσουμε κριτική. Οι πρόσφατες μελέτες δεν λαμβάνονται υπόψη, λαμβάνεστε σε κάποια, βασίζεται σε κάποια στοιχεία που δεν είναι βάσιμα, δεν είναι τεκμηριωμένα, δεν δημοσιεύετε τις μελέτες σε επιστημονικά έντυπα δεν λαμβάνεται υπόψη αυτά που αναφέρουν άλλες μελέτες και αυτό που είπε και η συνάδελφος Ροτ Μπέρεντ ε, στην ερώτηση της. Ουσιαστικά λοιπόν επαναλαμβάνω πρόκειται για ένα σκάνδαλο. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε η κυρία Λιωτάρ ή η κυρία Λεπάζ. Πέντε αποδείξεις δεν λαμβάνονται υπόψη ενώ ζούμε σε μια Ευρώπη που διακατέχεται από φόβο, από απάτες στον τομέα των τροφίμων, κάτι που έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των τροφίμων. Δεν μπορείτε εσείς σαν αρχή υπεύθυνη της ασφάλειας των τροφίμων να μην λάβετε υπόψη αυτό το φόβο οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται προστασία. Ε, βεβαίως, εδώ υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα. Και οι μελέτες, οι οποίες ε, υπαγορεύονται από βιομηχάνους, χωρίς απολύτως κανέναν ενδιασμό, θα πρέπει να αγνοηθούν, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Φίλα Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλισης των Τροφίμων για την παρουσία που μας έκανε. Θα ήθελα να μιλήσουμε για δόση ασπαρτάμις, όχι για ασπαρτάμι γενικά και αόριστα. Όλες οι μελέτες γίνονται με βάση συγκεκριμένε δόσεις. Όλοι οι τοξικολόγοι ε, γνωρίζουν πως ε, το θέμα δεν είναι η δραστική ουσία αλλά η δόση ακόμα και με νερό που είναι απόλυτα υγιεινό συστατικό κανείς μπορεί να πεθάνει αν το πάρει σε πολύ μεγάλες ποσότητες ε, γίνεται λόγος επίσης για σύγκρουση συμφερόντων όμως όταν βγήκαν οι μελέτες κατά της ασπαρτάμης και πάλι είχε γίνει λόγος για σύγκρουση συμφερόντων και πιο συγκεκριμένα για ένα για συμφέροντα ενός κατασκευαστή άλλη γλυκαντική ουσία πιο ακριβή από την ασπαρτάμ που θα μπορούσε όμως να την υποκαταστήσει. Εγώ εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Ασφάλιστων Τροφίμων ε, γιατί, ε, γιατί την πληρώνουμε αν δεν την εμπιστευόμαστε. Ας την καταργήσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω με τι δόσεις έγιναν οι μελέτες, οι δοκιμές και οι μεν και οι δε και οι πέρι και οι κατά της ασπαρτάμης. Ε, αν έγιναν με 40 μιλιγράμμ ανά κιλό ε, και βγήκε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αρνητικό για τον οργανισμό, δεν βλάπτει, τότε θα πρέπει να το πιστέψουμε. Um, Ευχαριστώ. Λέει η κυρία Γκέλλη. Εδώ έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, κάτι το οποίο δεν και τόσο συνείδηστο. Εάν θέλετε να μάθετε για τα διακυβευόμενα συμφέροντα των μελών του πάνελ, να, ρίξτε μια πια τώρα. Και αν έχετε κάποιο είδου ένσταση για τα συμφέροντα και τις συγκρούσεις των συμφερόντων, τότε αυτό θα πρέπει να δηλώνεται πριν τη συνεδρίαση όπου λέει ο καθένας ό,τι να είναι. Δεν είναι επαγγελματικό αυτό. Είναι, είναι συκοφαντικό. Να το λέτε όταν έχετε κάποιο πρόβλημα. Κοιτάξτε καλύτερα. Πώς εμπλέκονται και τι κάνουν. Ο τρόπος που εκφράζετε τις αμφιβολίες σας προσβάλλει την Επιτροπή. Αυτό ήθελα να πω. για τον είχα μιλήσει για Μακρόν και είχα επικρίνει την ΕΦΣΑ γιατί δεν έλαβε υπόψη όλες τις μελέτες και γιατί δεν έλαβε υπόψη κάποιες μελέτες που διαφωνούσαν με την ίδια την Και ε, τότε μου είχαν, με είχαν επικρίνει. Δεν σας αρέσει η Ασπαρτάμ και επιτρέψτε στην ΕΦΣΑ. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, εκτίθεστε γιατί αυτό είναι παράλογο. Κοιτάξτε καλύτερα γύρω τι γίνεται στον κόσμο. Μας παρουσίασε η ΕΦΣΑ τα στοιχεία που υπάρχουν. Σύμφωνο με την κυρία Αγίουσο. Χθες σα εξέπληξα κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ενημερώσω ότι πολλές φορές έχω επικρινή την Εύσα εδώ στη συνεργασία της Επιτροπής μας. Και ούτε με πληρώνει κάποια βιομηχανία, ούτε έχω κάποιον άλλο λόγο. Απλώς προσπαθώ για όλα αυτά να έχω την κοινή λογική. Κάτι το οποίο δεν το διπίστωσα σήμερα να πρέτανε. Και ρωτώ, πρόκειται για την πρώτη πανεξιολόγηση, σύμφωνα με όσο διαβάζω. Πότε θα γίνει η επόμενη επανεξιολόγηση και πόσες θα γίνουν. Αυτή είναι η ερώτηση που θέλω να θέσω. Ευχαριστώ πολύ. Κρατήσατε και το χρόνο ομιλία σα και εσείς έχετε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να συμφωνήσω με την κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ την Άτια την εργασία της. Και όλοι αυτοί που αμφισβητούν και μιλάνε για σκάνδαλο, να μας πούνε που βασίζονται. Δεν μπορεί όλα να είναι λάθη, κυρίως άμα δεν πετύχετε αυτό που πολιτικά θα θέλατε να πετύχετε. Δεν σας βολεύει το αποτέλεσμα των μελετών, άρα μιλάτε για σκάνδαλο. Η κυρία Γκέρλινγκ έχει δίκιο. Δεν το θεωρώ καθόλου σωστό. Δεν μας τιμά αυτό που κάνουμε εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Υπάρχουν επιστημονικές ε, μέθοδοι και υπάρχει τρόπος ε, αμφισβήτησης, ο οποίος πρέπει επίσης να είναι επιστημονικός. Δεν μπορούμε τώρα ξαφνικά επειδή δεν θέλουμε να περάσει κάτι και επειδή δεν μας βολεύει το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας να ε, λέμε ότι υπάρχουν πιέσεις και ότι φταίει η βιομηχανία, ο κλάδος, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες οι οποίοι χρηματοδότησαν και υπαγόρευσαν αυτές τις μελέτες. Δεν πρέπει να είμαστε λοιπόν τόσο υπερβολικοί γιατί ουσιαστικά δεν μπορούμε να ζητάμε κάθε φορά αυτό που πολιτικά μας βολεύει να στηρίζεται και από τους επιστήμονες. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί γιατί εδώ αμφισβητούμε μία αρχή και ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές ομάδες πίεσης που θα είναι πολύ ευτυχείς αν αυτή η αρχή πάψει να υπάρχει. Λοιπόν, το θέμα είναι η περιεκτικότητα όντως της ασπαρτάμης στα τρόφιμα. Η κυρία Γιώργο έχει δίκιο, είναι θέμα δόσης, όλα μπορεί να είναι δηλητήριο, αν η δόση στην οποία τα πάρουμε είναι υπερβολική ή δεν είναι αυτή που πρέπει. Ευχαριστώ πολύ και εσείς κρατήσατε, τηρήσατε το χρόνο ομιλία σας. you mentioned uh, Μιλήσατε για τον καρκίνο, αλλά μιλήσατε και για τις μελέτες για τα έμβρια. Γενικά όμως, τι, ε, ποια είναι η άποψή σας για τις ε, ορμονικές διαταράξεις. Δεύτερον, γιατί συμπεραίνεται ότι είναι απόλυτα ασφαλής. Οκ, okay, εντάξει λέτε είναι απόλυτα ασφαλής, αλλά γιατί δεν λέτε ε, αν είναι πιο ασφαλής ή λιγότερο ασφαλής από άλλες, ε, άλλες, άλλες εναλλακτικές γλυκαντικές ουσίες. Και βέβαια ε, έχω την διάποψη με τους υπόλοιπους και για το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Ε, ακόμα και το πώς είχε εγκριθεί η Ασπαρτάνη στις ΟΠΑ ήταν πολύ άσχημες οι διαδικασίες. Τελειώνοντας θα δώσουμε το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλής Τροφίμων. Έχουμε λίγα λεπτά. Εντάξει, έχουμε ακόμα λίγα λεπτά μέχρι τις ε, και 20. Είναι και 20, συγγνώμη. ευχαριστώ. Να σα πω κάποιε γενικέ παρατηρήσεις και οι συνάδελφοι μπορούν να συμπληρώσουν τα πιο λεπτομερή ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τη σύγκρουση των συμφερόντων, πρέπει να σας πω ότι το ελεγκτικό συνέδριο προέβη στον έλεγχο τη ΕΦΣΑ το 2007 και διαπίστωσε ότι η ΕΦΣΑ είναι από τις πιο προχωρημένες και ε, εντάξει υπηρεσίες όσον αφορά τη σύγκρουση συμφωνών. Γιατί υπήρχαν κάποιοι κανόνε παλαιότερα το 2002 που όντω ε, εμπόδιζαν τα, τα, τα πάνελ τη ομάδα εργασία και γι' αυτό και σα τονίζω ότι πρόσφατα ο διαμεσολαβητή ε, συνέταξε μια έκθεση για συγκεκριμένη περίπτωση και εκεί πέρα βεβαίωσε ότι η ΕΦΣΑ τηρεί τι προβληπόμενε διαδικασίε και με ένα νέο σύστημα τώρα γίνεται η επαλήθευση φαραγίζουν περισσότερο τη διαδικασία αυτή κλπ. Είχαμε κάποιες ε, συστάσεις τις οποίες και υλοποιήσαμε. Πρόχουν και πέραν της πενταετίας. Αλλού όμως υπάρχει πενταετία, αλλού προβλέπεται δεκαετία. Αυτό που χρειάζεται είναι υπάρχει συνέπεια. Εμείς θα ακολουθήσουμε τις χαμηλές γραμμές επράλεξης επιτροπής και αν τελικά προκύψουν κάποιες πρωτοβουλίες, θα τις εφαρμόσουμε αμέσως. Εάν έχουμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα για το ζήτημα το οποίο έθιξε η κυρία Μακάβαν, η κυρία Χέμπνερ, η συνάδελφος, θα μπορούσε να απαντήσει στην κυρία Μακάβαν. Ρωτήσατε κάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά συμφέροντα των ε, εμπειρογνωμόνων. Όπως είπατε σωστά, όλα αυτά δηλώνονται στην ετησία του οικονομικών συμφερόντων που είναι προσβάσιμα. Όλα αυτά ισχύουν σύμφωνα με τους του 2007 και αξιολογούνται και επανεξιολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες του 2012. Οπότε και οι εμπειρογνώμονες σαν συνέπεια παρετήθηκαν από αυτό το οποίο ε, προκαλούσε σύγκρουση συμφερόντων ή δεν λάμβαναν μέρο στο συγκεκριμένο πάνελ που δημιούργησε το πρόβλημα. Μα είπατε όμω αν υπάρχει εδώ κάποια σχέση με ε, την βιομηχανία των γλυκαντικών ουσιών. Θα μπορούσατε να μα εξηγήσετε τι εννοείται, αλλά πρέπει να σα πω ότι είχαμε κάποιον συνάδελφο που είχε λάβει μέρο σε κάποια επιτροπή ε, θα βράδυ κάποιου ε, επιστήμονε που ασχολούνται με την ασπαρτάμι, αλλά το 2009 πριν αρχίσει η ομάδα εργασία ε, ήταν αυτό, γιατί άρχισε το πάνη το 2012. Επίση, ε, είχαν συμμετάσχει σε κάποιο συμπόσιο όπου ήταν σπόνσορ Coca-Cola και δώσανε το 2009 κάποια διάλεξη για τις γλυκές ουσίες, αλλά αυτό ήταν πολύ πολύ καιρό πριν αρχίσει η δουλειά για την Ασπαρτάμι. Έχουμε ακόμα ένα λεπτάκι. Όσον αφορά τα δεδομένα, τη βιομηχανία, Αλήθεια είναι ότι η βιομηχανία συλλέγει τα δεδομένα και φτιάχνει αυτές τις μελέτες. Και είναι αλήθεια ότι και σε αυτή την περίπτωση συνέβαλε η βιομηχανία που συλλέξαμε εμείς τα στοιχεία. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικέ αυτές τις πληροφορίες. Αν θέλετε άλλο σύστημα, εντάξει, εμάς δεν μας πειράζει. Αλλά όσο ισχύει αυτό το σύστημα, τι να κάνουμε. Δεν ευνοούμε κανένα εις βάρος άλλου. Υπάρχουν κριτήρια και δεν καθόμαστε να μετρήσουμε το επιχείρημα της μιας της άλλης πλευράς. Προσπαθούμε απλώς να τηρήσουμε τα στάνταρ, τα ποιοτικά που υπάρχουν σε σχέση με τις μελέτες. είπε Και όπως σας είπα στην αρχή από αυτού, εμείς έχουμε μία ολόκληρη σειρά μελετών και καλύπτουμε στην εκθέση όλα αυτά τα οποία είπαμε στην εισήγησή μας. Καλύπτω αυτές τις μελέτες τώρα αν θέλετε βέβαια πιο επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις. Αυτό δεν μπορεί να είναι σαν λεπτό, θα σας τα πει ο συνάδελφος ένα λεπτό έχετε. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Regarding the criteria uh, for the studies, these... Όσον αφορά τα κριτήρια επί των οποίων βασίζονται αυτές οι μελέτες, είναι κρυστάλλινα. Το είπαμε στο παράρτημα της μελέτης για την Ασπαρτάνη. Είναι πολύ αυστηρά. Πώς συνελέγησαν τα δεδομένα, η τεκμηρίωση, τι γίνεται με τη συλλογή των δεδομένων, πώς ε, ερμηνεύεται ούτως η μελέτη, όλα αυτά περιγράφονται. Και αυτό ισχύει και για τις αρνητικές για να σπαρτάνε οι μελέτες και για τις θετικές. Τα στάνταρ τα οποία ακολουθούμε είναι παγκοσμίω αναγνωρισμένα. Επίσης σας τονίζω ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ακριβώς τα ίδια. Και για τις αρνητικές και για τις θετικές μελέτες σε σχέση με τις επιπτώσεις επί της υγείας. Καμία δεσμής διάκριση δεν έγινε. Τώρα το τελευταίο. Η θηρασύνη, τα ενδοκρινολογικά, όλα αυτά τα είδαμε. Όμως, θεασίνη και τα υπόλοιπα μηνοξέα δεν γνωρίζουν μια άλλη μεταβολία. σε ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν απαντήσαμε σε όλα τα ανοιχτά ερωτήματα, αλλά έτσι και αλλιώς ε, το σημείο αυτό θα μας ξαναπασχολήσει. Στο 24 σημείο της ημερήσιας διάταξης έχουμε τις ημερομηνίες για την προσεχή συνεδρίαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου στέλνει το λόγο. Okay, thank you Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας εξηγήσω τις συνθήκες που αφορούν την υιοθέτηση του κανονισμού προέλευσης. Ε, στείλετε και μια επιστολή στον Επιτρόπο Τσιόλος και στον Επιτρόπο Μπόργκ ε, όπου φράζετε τις ανησυχίες, ε, τις σας για τον περισμένο χρόνο που δίδεται στο Κοινοβούλιο για να εξετάσει τα μέτρα που προτείνονται. Το προτινόμενο κείμενο αναρτήθηκε, στο, καταχωρίστηκε στις 26 Νοεμβρίου ε, και η, ψηφοφορία έγινε στις 5 Νοεμβρίου. Ε, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα ε, εξαιτία ενός δυσάριστου διοικητικού προβλήματος και εξαιτία των χρονικών περιορισμών που έχει η Κομισιόν που θα πρέπει να υιοθετήσει τους κανόνες αυτούς μέχρι τέλο του χρόνου. Επί τώρα, Πρόεδρε. Η προετοιμασία αυτού του εφαρμοστικού κανονισμού ε, ε, έρχεται κατόπιν μελέτης που είναι διαθέσιμη. Στη δεύτερη φάση οι υπηρεσίες κομισιών έκαναν και μια μελέτη επιπτώσεων σε ό,τι αφορά τις διάφορες δυνατότητες που ε, υφίσταντο με βάση την βασική πράξη. Ε, αποδείχθηκε ότι οι, πιο θετικές ήταν οι, επιλογές που Πρώτον, το κράτος μέλος διατηρεί το γεωγραφικό του επίπεδο και δεύτερον, συστήματα για τον καθορισμό ε, του, ε, της, των κανόνων προέλευσης ε, με βάση την γέννηση του ζώου, του μόσχου. Οι δύο μελέτες συμπρογνωμών ήταν πολύ λεπτομερείς ε, και προσπαθήσαμε τα πορίσματά τους να τα εντάξουμε στο κείμενό μας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου, των νέων κανόνων, του νέου κανονισμού είναι πιστεύουμε ότι αποτελεί ο κανονισμός ομοιόμορφος και σαφής κανόνας για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπεριλαμβάνει ε, την τους διατάξεις χνηλασιμότητας που προσδιορίζουν ε, την ε, πρόληψη στην καταγωγή και καθιστούν τους κανόνες αξιόπιστους. Θέτει ως baseline για το κρέας το οποίο καλύπτεται την ένδειξη σφαγής και και τροφής ε, έτσι ώστε ε, να αποδεικνύεται ότι ε, το ζώο έχει περάσει ένα μεγάλο τμήμα της ζωής του στο συγκεκριμένο κράτος από το οποίο θεωρείται ότι κατάγεται. τώρα, οι αναφορές στην σφαγή ή στην ε, κτροφή μπορούν να αντικατασταθούν από την ένδειξη προέλευσης ε, μόνο αν το ζώο έχει γεννηθεί, μεγαλώσει και ε, σφαγεί εκεί και υπό την προπόθεση θα συμφωνήσουν και οι εθνικές, αντίστοιχες εθνικές αρχές. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα οι εμπορευόμενοι να συμπληρώσουν τις υποχρεωτικές ενδείξεις με πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες υπό την προπόθεση ότι αυτό είναι συμβατό με τους εφαρμοστέους κανόνες. Αυτά σε ό,τι αφορά το, την ουσία του κανονισμού. Στο τέλος της διαδικασίας συζήτηση με τα κράτη-μέλη, η ψηφοφορία στις 5 Νοεμβρίου απέδειξε ότι υφίσταται μια σαφής ε, ειδική πλειοψηφία υπέρ της πρότασης. Ε, και οι οργανώσεις των καταναλωτών και οι οργανώσεις της, ε, του κλάδου είδαν θετικά τους νέους κανόνες. Η συζήτηση αυτών των εφαρμοστικών κανόνων ήταν μια περίπλοκη και σύνθετη διαδικασία. Ε, το τελικό αποτέλεσμα ήταν καλό συμβασμό και θα βοηθήσει του κατανοητέ να κάνουν ε, τι ε, επιλογέ του πληροφορημένοι. Βέβαια, ε, δεδομένη τη βιασύνη εξαιτία των προθεσμιών, υπήρχε μόνο μία εβδομάδα μεταξύ της κοινοποίηση του κειμένου σε εσά και της προφορίας στην Επιτροπή. Λυπάμαι γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι ε, σας υπόσχομαι πως θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σόμερ. Κοιτάξτε, αυτή η επιταχυμένη διαδικασία δεν είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος. Βεβαίως μπορούμε εμείς να εκφράσουμε διαφορετικές ε, απόψεις και επιχειρήματα, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ε, κανονική διαδικασία και χρόνος επεξεργασίας. Τώρα, ποιο είναι το κόστος όλης αυτής της ιστορίας. Πάρα πολύ περίπλοκο το βρίσκω το σύστημα και αυτό ήθελα να πω στην Επιτροπή. Και πραγματικά αμφισβητώ και το κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί. Τι να σας πω, δεν μας έχετε στείλει τίποτα, ξαφνικά πραγματικά έρχεται όλο αυτό το πακέτο και θέλω να σας πω ότι εξοργίζομαι. Κοιτάξτε, ήταν ξεκάθαρο ότι εμείς σκεφτόμασταν κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει με το βόλιο κρέας. Εδώ μας κάνετε μια τελείως διαφορετική πρόταση από αυτό που ισχύει στο νο κρέας, όπου λέμε έχει εκτραφεί, έχει σφαγιαστεί την χώρα. Σας ρωτώ λοιπόν τι έγινε, γιατί εδώ παραδείγματος χάρη να υπάρχουν τρία διαφορετικά μέρη, ε, τι κάνετε, πώς το συμπεριλαμβάνετε στις ενδείξεις επίσης όσον αφορά τις ε, τιμές. Εδώ αυτές οι μη ρεαλιστικές αυξήσεις τιμών, αυτή η εναλλακτική λύση που προτείνεται ουσιαστικά δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση των τριών τόπων. Ναι, μπορεί να μας πείτε βέβαια ότι είναι καλύτερο να έχουμε αυτό από το μηδέν και έτσι θα πετύχουμε και την ειδική πλειοψηφία. Αλλά πώς το λαμβάνετε υπόψη. Εμείς πραγματικά εκνευριζόμαστε και δεν είμαι ο μόνος γιατί δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα σχόλιά μας. Και επαναλαμβάνω αυτό που προτείνει εδώ η Επιτροπή δεν συμπεριλαμβάνει καν τις ε, βασικές μας διαμαρτυρίες όπως αυτά που σας είπα για τους τρεις τόπους που δεν λαμβάνονται υπόψη γεννήθηκε, εξετράφει και έχει σφαγιαστεί παραδείγματος χάρη. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Κυρία Μακέβεν. Ευχαριστώ. Ο, μιλάω εξ ονόματος της ε, Evans. Το θέμα δεν είναι για δύο ή τρία. Για το βόλιο κρέας έχουμε τις τρεις δυνατότητες. Στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει αυτού του είδου η σήμανση για το βόλιο κρέας. Γιατί δεν κάνουμε το ίδιο κι εμείς. Γιατί δεν ισχύουν εδώ τα ίδια πρότυπα. Ας κοιτάξουμε μια φορά το τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού γιατί βλέπετε ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους αδυναμίες και δυνατότητες θα τις εκμεταλλευτούν οι επιτίδοι. Και θα πούνε ότι η τελική επεξεργασία, παραδείγματο χάρη, έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε εδώ. Γιατί δεν είμαστε ξεκάθαροι να ξέρουν οι άνθρωποι τι αγοράζουν και τι τρώνε. Σήμερα ξέρετε ότι πάρα πολλά σούπερ μάρκετ ήδη ε, έχουν τέτοιες ενδείξεις, γιατί το ζητάει ο καταναλωτής. Γίνεται, είναι δυνατό να γίνει και ήδη συμβαίνει. Γιατί λοιπόν να μην το απαιτήσουμε. Ας κάνετε μία φορά κάτι σωστό. Ναι, εγώ θα ήθελα να πάρω το λόγο, λέει, κυρία Σόμερ, γιατί κάποια τμήματα του Κοινοβουλίου, μία μειοψηφία, είχε ζητήσει αυτή τη διαδικασία με τρεις ε, δυνατότητες, τρία επίπεδα και τελικά έγινε μια εξέταση αυτού του συστήματος. Το είχε ζητήσει η Επιτροπή. Αυτές, αυτές οι τρεις βαθμίδες προέλευσης αν θέλετε δεν είναι κάτι το αυτονόητο. Εμείς είχαμε ζητήσει αν ναι ή όχι αυτό μπορεί να γίνει, αν είναι υλοποιήσιμο. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτής της ε, εξέτασης ήταν ότι δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ο καταναλωτής δεν θα υποφεληθεί τόσο πολύ. Το θέμα τώρα της προστασίας των ζώων. Αυτό είναι εδώ που ζητάμε ή η προστασία του καταναλωτή. Δεν ξέρω ας είναι ξεκάθαρος ο σκοπός. Γιατί παραδείγματος χάρη η μεταφορά των ζώων, ο τρόπος ε, σφαγιασμού, το θέμα της προστασίας της ευημερίας των ζώων είναι άλλο θέμα και φυσικά και θα πρέπει να το λάβει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή. Αλλά το θέμα τώρα της προστασίας του καταναλωτή, της ασφάλειας των τροφίμων, ας τοποθετηθούμε σωστά, γιατί άκουσα πολύ προσεκτικά τι είπαν οι συνάδελφοι και αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι οι πληροφορίες και οι οδηγίες. Όχι, αυτό που λέτε δεν ισχύει, λέει ο Πρόεδρος. Αυτή η τοποθέτηση ήταν τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις τρεις βαθμίδες. σήμανση με τρεις βαθμίδες. Ναι, αλλά κοιτάξτε, το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης δεν ήταν αυτό. Επαναλαμβάνω, λέει ο Πρόεδρος, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν αυτή. Σήμανση με τρεις διαφορετικές βαθμίδες. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι σωστά, είναι λάθος και δεν είναι και ειλικρινής παρουσίαση των γεγονότων. Η διαπραγμάτευση ήταν ένα θέμα. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι αυτή που σας λέω. Είπατε η θέση του Κοινοβουλίου. Αυτό είπατε. Και αυτό είναι λάθος. Αυτό που ε, ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν είναι αυτό που λέτε. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι λάθος αυτό που λέτε. Η θέση ήταν οι τρεις βαθμίδες. Μα κοιτάξτε, δεν είναι αυτό το ουσιαστικό. Εμείς συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, μετά τη διαπραγμάτευση γίνεται τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Ναι ή όχι. Εάν προηγουμένως το Κοινοβούλιο είχε μια άλλη θέση, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, ένα άλλο προηγούμενο στάδιο, είναι άλλο θέμα. Τελικά η θέση του Κοινοβουλίου είναι το αποτέλεσμα της διαβούλευσης, της συμβιβαστικής αυτής ε, διαπραγμάτευσης. Αυτή γίνεται στο τέλος η θέση ε, του Κοινοβουλίου. Δεν καταλαβαίνω. Η αρχική θέση του Κοινοβουλίου με την οποία μπήκαμε στη διαπραγμάτευση ήταν σήμανση τριών βαθμίδων. Αυτό είχαμε συμφωνήσει. Και μετά έγινε διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Ωραία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνετε ότι η Κομισιόν εργάζεται επί του κειμένου που υιοθετήθηκε τελικά. Και λέει ακριβώς αυτό, άρθρο 26 παράγραφος 9. Μεταξύ άλλων θα εξετάσει τις δυνατότητες έκφρασης των κανόνων προέλευσης με βάση τα ακόλουθα σημαντικά σημεία. Σημείο γέννηση, σημείο εκτροφής, σημείο σφαγής. Οπότε το νομικό κείμενο έχει δυνατότητες, εναλλακτικές δυνατότητες. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, έκαν, κάναμε μια μελέτη επιπτώσεων και λάβαμε υπόψη τα ενδιαφέροντα όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών βέβαια, αλλά όχι μόνο των καταναλωτών και των εμπορευομένων. Ένα άλλο Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι το κόστος. Το εκτιμόμενο κόστος αυτού του κανονισμού είναι 1 έως 2% της αξίας του ζώου. Εκεί το εκτιμήσαμε. Υπάρχει, λόγη, υπάρχει λόγος για τον οποίο δεν είναι δυνατή η ανεγγραφή του γεννήθηκε στην. Ε, ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι οι κύκλοι παραγωγής για αυτά τα ζώα, ε, χείρους, ε, ε, για τα άλλα ζώα, δηλαδή χείρους, κοτόπουλα κλπ. είναι πολύ πιο μικρής διάρκειας. Για παράδειγμα, το τόπος γέννησης για τα κοτόπουλα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους καταναλωτές. Στο σύστημα ταυτοποίησης των ζώων αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται η χνηλασιμότητα του τόπου γέννησης για όλα αυτά τα ζώα. Ε, δεν δίνεται μάλλον αυτή η δυνατότητα. Η επιβολή αυτών των όρων θα αποτελούσε πρόσθετο κόστος, το οποίο η μελέτη επιπτώσεων δεν θεώρησε δικαιολογημένο. Επίσης, έγινε ερώτηση για τον κοιμά. Ο κανονισμός προβλέπει την ίδια baseline για όλα τα προϊόντα και για αυτά τα προϊόντα όπως και για τα υπόλοιπα είδη κρέατος. Όμως η αλήθεια είναι πως ε, η ε, παρασκευαστές των ε, κοιμά ε, αναμειγνύουν ομόκριας από διάφορα ζώα. Οπότε θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους εμπορευομένους να, θεωρήσουν, να δώσουν ως ένδειξη καταγωγής, προέλευση μάλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ως απάντηση των βασικών ανησυχιών. Einmal kurz eine Nachfrage bei Karl Schlüter, bitte. Karl Schlüter, μια σύντομη ερώτηση. Σε ποια μέρη τι αναφέρεστε όταν λέτε ότι οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται το που γεννήθηκαν τα κοτόπουλα και δεύτερον, ποιες οργανώσεις καταναλωτών ικανοποιήθηκαν για το ότι αναφέρετε δύο τόπους αντί για τρεις. Είπατε ότι ήσαν ικανοποιημένοι. Τι εννοείτε. Δυστυχώ μετά από αυτή την απάντηση πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κύριε Σλούτερ, δεν λέω ότι ήταν ικανοποιημένοι. Είπα ότι προσπαθήσαμε να βρούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων θέσεων, μεταξύ των παραγωγών και όλων των υπόλοιπων φορέων. Και τελικά είπαμε ότι το ενδιαφέρον του τόπου γέννησης, η προσθέμενη αξία αυτής της ένδειξης ήταν ε, λιγότερο σημαντική. Ευχαριστώ πολύ. Θα συναντηθούμε της 9 ε, Ιανουαρίου, κατόπιν θα ψηφίσουμε στις 23 Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ όλους τους ε, συνεργάτες και τους διερμηνείς. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να συνεδριάσουμε εδώ και σας εύχομαι σε όλους καλές ε, γιορτές, καλή χρονιά και καλή αντάμωση τον Ιανουάριο.